I think we can start. Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κυρίσω την έναρξη συνεδρία της Επιτροπής μας. Ε, μπορεί να εγκριθεί η μερίσια διάταξη, αν δεν διαφωνεί κανείς, υποθέτω. Ωραία, εγκρίνεται. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, μπορούμε να εγκρίνουμε και τα πρακτικά της 26 Σεπτεμβρίου και 11 και 11 Οκτωβρίου. Ωραία, και εδώ δεν έχουμε αντίρρηση. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Μέχρι τώρα τίποτα. Και πάμε στο 4 αμέσως. Ε, το δέσμη ε, μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Τρία θέματα είναι η διάνοιξη των αγορών ε, για τις επιβατικές μεταφορές, η διαχείριση των δικτύων και οι λογαριασμοί των σιδηροδρόμων. Πρέπει να σας πω κάτι διαδικαστικό στην αρχή. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου στις 27 Οκτωβρίου στην Ολομέλεια κοινοποίησε τις θέσεις ε, του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για τα τρία θέματα. Σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 2 του κανονισμού μας προβλέπονται τα εξή και παραθέτω. Η θέση του Συμβουλίου εγγράφεται ως πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίας της ε, Καθήλυνα Αρμόδιας Επιτροπής ε, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης. Τέλος παράθεσης, εμείς είμαστε αρμόδιοι επί της και κοινοποιώ και εγώ ότι έχει φτάσει η κοινή θέση, οι κοινέ θέσει του Συμβουλίου και αρχίζει να μετράει η δεύτερη ανάγνωση και επίσημα και τυπικά για την νομοθεσία. Οι συγκητέ ήδη αύριο θα καταθέσουν τι συστάσει τους για τη δεύτερη ανάγνωση. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου εδώ στην Επιτροπή, ενώ στην Ολομέλεια το Δεκέμβρη. πάμε στο σημείο 5 στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη, έκθεση πρωτοβουλίας δική μας είναι, εισηγητής ο Πάβελ Τέλιτσκα και του δίνω μέσα στο λόγο. Ε, Πρόεδρε, συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, καλημέρα και ευχαριστώ για το λόγο. Πρώτα απ' όλα να επαναλάβω κάτι που έχω πει και προηγουμένω στην Επιτροπή μας. Ότι μαζί με τους Κιώδης έχουμε συμφωνήσει σε κάποιες βασικές αρχές επί των οποίων θα θέλαμε να στριχθούμε για τη στατική μας περιοχή Πρώτα απ' όλα, καταλαβαίνουμε όλοι, ευτυχώ ότι πρέπει να σχεδιάσουμε στρατηγική, ώστε να συμπεριλάβουμε όσα υπάρχουν ήδη στην νομοθεσία, όσα θέλουμε να υλοποιηθούν και να δούμε τι δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Όμω πρέπει να έχουμε μια εικόνα κάπω ε, διορατική για το μέλλον διορατικότητα μάλλον. Θα πρέπει να κοιτάξουμε την αεροπλοεία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας για τις Συγκοινωνίες και θα πρέπει να τονίσουμε και να αντικατοπτρίσουμε κάποια ζητήματα που είναι κέρια σε αυτό το πλαίσιο αλλά που μπορεί να επηρεάζονται και από τι αρμοδιότητε άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών του Κοινοβουλίου. Θέλουμε να είμαστε αρκετά συγκεκριμένοι Επίσης να τονίσω ότι μεταξύ των βασικών στόχων ήταν να δούμε το θέμα της ε, διασύνδεσης για το μέλλον, καθώς και της, ε, του συνδυασμού πολλών διαφορετικών τρόπων συγκοινωνιών. Για την ασφάλεια, επίσης θα πρέπει να λάβουμε την μέρημνα, καθώς η δαπάνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα θέμα που θα επηρεάσει εδώ. Για τη στατική μας περιοπλοίας, με τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί πρέπει να πούμε ότι γίνεται σεβαστή εσωτερική συλλογιστική την οποία διατηρούμε και στις τροπολογίες και μπορούμε να εισάγουμε κάποια σημεία τα οποία είναι σημεία κλειδιά για μας, τις πολιτικές μας ομάδες. Έχω ένα συνάδελφο που με προσπερνάει και μου καταστρέφει λίγο τα χαρτιά μου. Είναι ο κύριος Δίλερ, μπορούμε να συμφωνήσουμε και να το δεχτούμε. Ε, είναι ψηλό τι να κάνουμε. Ε, εδώ λοιπόν υπάρχει μια εσωτερική δομή και συλλογιστική και γι' αυτό να εκφράσω την εκτίμησή μου προς τους συναδέλφους. Σε αυτό το πλαίσιο να αναφέρω ότι με τα χαράς θα συνεργαστώ με τους συναδέλφους. Ξέρω ότι είναι μια μορφή κλασικής ευγένειας να ευχαριστεί στους τους κοιόδες όμως πραγματικά εδώ έχω συναδέλφους που είναι ιδιαίτερα επαείοντας στο συγκεκριμένο τομέα, ε, με ιδιαίτερη το, ισορρο, ισορροπή εκπροσώπηση των φίλων, είναι όλοι επαγγελματίε του χώρου και συνάδελφοι να πω ότι πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε επιτυχώς στην όλη διαδικασία εφόσον έχουμε τροπολογίες που θα μας οδηγήσουν σε ικανοποιητικού συμβιβασμούς. Έχουμε ακόμη δύο συνεδριάσεις. Μία έγινε μόλις χθε με τους Κιώδης. Ελπίζω ότι θα καλύψουμε και άλλο μέρος της ύλη μας και θα πετύχουμε μια συμφωνία τουλάχιστον μεταξύ μου για κάποια ζητήματα που θα πρέπει να επιληθούν είναι το συν Θα πρέπει λοιπόν να συνεννοηθούμε με τις πολιτικές μας ομάδες. Νομίζω όμως ότι βαθμός αφοσίωσης όλων και διάθεσης να πετύχουμε είναι τόσο μεγάλος που ακόμα και αυτά τα πρέστατα σημεία δεν θα αποτελέσουν πρόβλημα. Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να περάσω ε, στην εξέταση των βασικών τροπολογιών, διότι τόνισα ποια είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν στην πρώτη συζήτηση. Θα ήθελα λοιπόν να σταματήσω σε αυτή τη φάση και θα ήθελα να ακούσω και τους Κιώδης και τα μέλη της Επιτροπής. Και αν χρειαστεί θα περάσω σε περισσότερες λεπτομέρειες όσο δεν στο τέλος της συζήτησης. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κλούν. good morning and, um, Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλημέρα σας. Ήθελα να ευχαριστήσω τον συναδελφό για την αρχική του έκθεση, η οποία ήταν πολύ καλή και στην οποία εν μέρει μπορέσαμε να συμφωνήσουμε και από όλε τι ομάδε, σωστά έχει ανακεφαλαιώσει την αίσθηση που επικρατεί σε όλε τι συνεδριάσει που είχαμε μεταξύ σκιωδών. Θετική διάθεση. Και υπάρχουν ακόμη κάποια ζητήματα αυτή τη στιγμή. Αλλά θα επιληθούν πιστεύω πώ οδεύουμε προ το τέρμα. Τα έχουμε συζητήσει ήδη στην Επιτροπή μα. Και ήθελα έτσι εξ αρχή να καταστήσω σαφέ ότι υπήρχε και γνωμοδότηση τη ΕΜΠΛ, τη Επιτροπή ΕΜΠΛ για την στρατηγική αεροπλοεία. Οπότε έχουμε εδώ να ασχοληθούμε μόνο με τα, καθή, τα κατεξοχήν ζητήματα αεροπλοεία, τα οποία διαφοροποιούν ε, λίγο τη δική μα δουλειά από αυτήν τη Επιτροπή ΕΜΠΛ. Εδώ θέλω να τονίσω την ανάγκη η Επιτροπή και τα κάτι μέλη να αναλάβουν δράση για ζητήματα όπω ο ενέο Ευρωπαϊκό Ουρανό, τα δικαιώματα των επιβατών, η νομοθεσία για τις κρίσεις αεροπλοείας, εδώ θέλουμε να προχωρήσει η αεροπλοεία, να γίνει πιο ανταγωνιστική και εσωτερικός, αφού προηγουμένως ε, τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας, σε εθνικό επίπεδο δούμε τα θέματα ανταγωνισμού, να περάσουμε και στη διεθνή διάσταση. Και σε αυτά που γίνονται με τους γειτονές μας. Υπάρχει μια ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι αυτά πρέπει να επιληθούν. Οι υπερπτήσεις Νομίζω δίνουμε μια καλύτερη κατεύθυνση από την αρχική έκθεση. Και φέρετε όλες οι πολιτικές ομάδες να έχουν ε, δείξει θετική διάθεση. Εναγνωρίζουμε την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών. Και υπάρχει ανάγκη να προχωρήσουμε και εδώ. Από τη στιγμή που συντάχθηκε η αρχική έκθεση, είχαμε στο Μορεάλ την ε, διάσκεψη της ΙΚΑΟ, οπότε και αυτό καλό να πηχηθεί στην έκθεση. Ο κύριος Τσαρνεύσκη ανέφερε το θέμα της ε, διασύνδεσης διαφορετικών ε, περιοχών μεταξύ τους Καλό θα ήταν λοιπόν να δούμε αυτό με τα κομβικά σημεία, τα hubs που μπορούν να δημιουργηθούν, την διασύνδεση διαφορετικών γραμμών μεταξύ του και κάποιε περιοχέ που δεν θέλουμε να παραμείνουν απομονωμένε. Διότι εξαρτώνται αποκλειστικά από την αεροπλοεία. Είναι σημαντικό και αυτό να αντικατοπτριστεί στην έκθεση. Συνολικά, σωστά αντικατοπτρίζονται οι συζητάσει που είχαμε προηγουμένω είναι λοιπόν θετική η αποτίμησή μα και χαιρόμαστε που υπάρχουν φιλοδοξίε για τον τομέα αεροπλοεία τη Ευρώπη. Όχι μόνο προ τι πτήσει, αλλά συνολικά για τι υποδομέ των αεροδρομίων, καθώ και την ε, αλυσίδα παροχή υπηρεσιών τη αεροπλοεία. Νομίζω θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας το Δεκέμβριο και μετά θα περάσει το θέμα την Ολομέλεια. Και πάλι να πω τη και να ευχαριστήσω τον κύριο Τσανέσκη για το ανοιχτό του πνεύμα και τον τρόπο που προείδρευσε σε όλε τι συναντήσει των σχεδόν από την αρχή, καθώ και όλου του συναδέλφου για την αφοσίωσή του. Θετική συνεισφορά όλων. Ευχαριστώ πολύ, κυρία ε, Νέσα Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή και κυρίως να τον ευχαριστήσω για την υπομονή που έδειξε και να πω πως ε, τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα και για το επίπεδο συνεργασίας που έχουμε πετύχει ε, μεταξύ μας οι σκιώδεις εισηγητές. Παρόλο που η δική του προσέγγιση ήταν μια στρατηγική για το μέλλον, πιστεύουμε πως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα στοιχεία τα οποία εφίστανται αυτή τη στιγμή και από τα οποία ξεκινάμε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να επιμείνουμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη μη αποδοχή της, του αθέμητου ανταγωνισμού από τρίτα κράτη και κυρίως για θέματα κρατικών ενισχύσεων, γιατί στην Ευρώπη ξέρετε πως δεν υπάρχουν πλέον. Αντίθετα όμως σε τρίτες χώρες ακόμα είναι ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Πρέπει να σας πω πως ε, για τα περιφερειακά αεροδρόμια και το πώς συνδέονται με τους μεγάλους κόμβους, εδώ δεν είναι μόνο η πολιτική εδαφική συνοχής, αλλά έχουμε και το δυναμικό κομμάτι που έχει να κάνει με το πώς μπορούν να συνδέονται περισσότερα αυτά τα αεροδρόμια για να ενισχυθεί το δυναμικό τους. Επίσης σας ευχαριστώ που έχετε συμπεριλάβει όχι μόνο τις υπερπόντιες περιοχές, αλλά και τα νησιά γιατί και εκεί αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα και μάλιστα εδώ υπάρχει και ένα στοιχείο ε, επιπλέον που είναι τα ορεινά νησιά που υπάρχουν ακόμα περισσότερα προβλήματα πρόσβασης στα αεροδρόμια τους. Κάποια στοιχεία πολύ σημαντικά για τα δικαιώματα των επιβατών είναι οι νέες τεχνολογίες που μπορούν να βελτιώσουν και να διευκολύνουν ε, και την πρόσβαση αλλά και το επίπεδο διαφάνειας ε, τη στιγμή που γίνεται η αγορά κάποιων ε, τουριστικών πακέτων. Όπως επίσης η ευελιξία. Να σας πω δε πως ο συμβιβασμός που πετύχατε, που νομίζω στηρίζεται από τις περισσότερες ομάδες, είναι ένα συμβιβασμό τον οποίο μπορούμε να δεχτούμε. Τέλος, υπάρχουν δύο σημεία τα οποία ακόμα είναι σε κρεμότητα. Ένα είναι η παράγραφος για τις κοινωνικές επιπτώσεις. Εμείς συμπεριλάβαμε πολλά κομμάτια που θεωρήσαμε σημαντικά, γιατί η Επίτροπος κυρία Μπούλτς είχε δεχθεί στην αρχή της θητείας της να φέρει ε, στο Κοινοβούλιο τουλάχιστον για καθένα από τους κλάδους ένα κοινωνικό πακέτο έτσι ώστε να φέρει μια ισορροπία μεταξύ των προβλημάτων ε, διαρροής ή μη ελκυστικότητας των κλάδων αυτών και αυτό συμπεριλαμβάνει και την αεροπλοεία για τους νέους εργαζόμενους, οπότε εκεί θέλουμε να δώσουμε κάποια συνέχεια. Επίσης, έχουμε ε, τους αυτοκινητοδρόμους των εθέρων, όπου εκεί ο εισηγητής για τα ανώτερα στρώματα αυτών των διαδρόμων δεν έχει πει κάτι το ιδιαίτερο. Νομίζω πρέπει να το συζητήσουμε με την ομάδα μας για να δούμε πώς μπορούμε να το δούμε, ε, να το θεωρήσουμε ως μια ε, δύο διαφυγής σε περιπτώσεις που αυτό χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τζακή Φώστερ είναι επόμενη και Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, ο οποίος από την αρχή όλων αυτών των συζητήσεων ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός. Όλα έχουν γίνει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η συνεργασία ήταν εξαιρετική. Όλοι εμείς οι σκιώδεις ε, κάναμε πάρα πολλές προσπάθειες έτσι ώστε να κάνουμε κι εμείς η δουλειά μας. Οπότε δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για όλα τα σημεία. Αν δούμε όμως την έκθεση ε, για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική, γιατί νομίζω ότι εδώ μιλάμε πια για στρατηγική, θα δούμε πως όλα τα κομβικά σημεία ε, στα οποία ο εισηγητής έχει σταθεί συμπεριλαμβάνονται. Και επίσης πρέπει να σας πω πως ο τρόπος με τον οποίο έχει διαστρωθεί είναι απλός, δεν είναι υπερβολικά ε, πομπόδης ο τρόπος που διατυπώσει το κείμενο και το έγγραφο αυτό έχει μεν 500 σελίδες, αλλά μπορώ να σας πω ότι τα όσα αναφέρει είναι τα κατάλληλα. Πολλές φορές βέβαια σε 25 σελίδες μπορούμε να πούμε τα ίδια με όσα λέμε σε 500. Τώρα για τις μεταφορές και για τη στρατηγική που προκύπτει από την ε, δική μας Επιτροπή πολύ σωστά ασχοληθήκαμε με τα κοινωνικά θέματα. Βεβαίως και θέλουμε να διασφαλίσουμε θέσεις εργασίας. Είναι ένας χώρος που μπορεί να φέρει ανάπτυξη Έχουμε το θέμα του περιβάλλοντος. Μην ξεχνάμε πως όταν συζητάμε τους ε, καθαρούς εθέρες, η αεροναυπηγική βιομηχανία, το κοινοβούλιο και άλλοι θεσμοί έχουν ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Έχουμε τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Όλα αυτά είναι θέματα που θα μας απασχολήσουν πολύ στο μέλλον και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σίγουροι πως αυτά θα λειτουργήσουν όταν όμως έχουμε την απαραίτητη πολιτική βούληση εμείς στα κράτη-μέλη. Και νομίζω πως κάποια κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή δεν επιδεικνύουν πως έχουν τη, τη βούληση να ενδυναμώσουν το δυναμικό μας και δεν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσει του 21ου αιώνα. Γιατί υπάρχει ένα μπλοκ κρατών που αυτή τη στιγμή έχουν εμπορικές σχέσεις με την υπόλοιπη ε, φίλιο, άρα λοιπόν θα πρέπει τα κράτη-μέλη να βάλουν το σημείο αναφορά, να τραβήξουν μια γραμμή και να δούμε τι πρέπει να πετύχουμε τώρα. Για την ασφάλεια, που είναι ένα θέμα στο οποίο έχουμε σταθεί και που γνωρίζετε κι εσείς, Πρόεδρε, πως είναι πολύ περίπλοκα τα συστήματα ασφάλειας για όσους περνάνε από τα αεροδρόμια και βεβαίως η ασφάλεια είναι σημαντική και είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε. Όμως, εκτός ότι είναι όλο και πιο δαπανηρή, νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε και πιο εξελιγμένους τρόπους για το πώς μπορούμε να το πετύχουμε, τουλάχιστον για τους ε, επιβάτες που ταξιδεύουν συχνά. Και είδαμε κάποια ε, πειράματα που έχουν γίνει στις ΗΠΑ για το free track, την ελεύθερη διέλευση, και να σκεφτούμε λιγάκι εκτός πεπατημένης για να δούμε πώς μπορούμε με την εμπειρία μας να βελτιώσουμε τα πράγματα έτσι ώστε να μην αποθαρρύνουμε όσους ταξιδεύουν για επαγγελματικά ταξίδια ή για διακοπές. Γενικά για τη συμφωνία χρειάζεται, χρειάζεται ανταγωνισμός και για την διασυνδεσιμότητα. Όπως είπε και η Τίτρη, είχαμε και εγώ πονήσει. Είμαι από την Ιρλανδία. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε το θέμα ε, των μικρών αεροδρομίων, το πώς αυτοί οι μικροί τόποι πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Θεωρώ λοιπόν πως η στρατηγική αυτή είναι πολύ ισορροπημένη και θα πρέπει να στηριχθεί από την ομάδα μου και σίγουρα θα στηρίξει σε μεγάλη της πλειοψηφία και αυτή η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Γενικότερα να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή για το πόσο αποτελεσματικά χειρίστηκε αυτό το φάκελο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κονέτσινα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις προτάσεις που κατέθεσε, για την προσέγγιση την οποία ακολούθησε. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητική η στάση του καθ' όλη τη διάρκεια των συναντήσεων και σεβάστηκε τις απόψεις μας. Βέβαια, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με όλα τα σημεία. Πρέπει να πω πως ε, μέσα στους βασικούς στόχους για τη στρατηγική αυτή Είπαμε πως σε όλες τις ε, συμφωνίες θα πρέπει να έχουμε τη βελτίωση της διασυνδεσιμότητας ως βασικό στοιχείο ε, γιατί βλέπω ότι εσείς βασίζετε πιο πολύ στις ανάγκες της αγοράς. Κάτι με το οποίο εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Εμείς τονίζουμε την ανάγκη που έχει ο καταναλωτής και όσοι δουλεύουν στην, ε, στον κλάδο της αεροπλοείας θα πρέπει αυτά να ληφθούν υπόψη πιο πολύ. Σεβόμαστε βέβαια την ε, έκθεσή σας κύριε Σίτα, αλλά δεν μπορούμε να την δεχτούμε γιατί πιστεύουμε πως θα πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του Ευρωπαίου πολίτη. Δηλαδή τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων στον ε, κλάδο της αεροπλοείας που είναι εξίσου σημαντικά για όλα τα κράτη-μέλη. Θα έπρεπε λοιπόν να τους προσφέρουμε τα εχέγγυα που θα τους επιτρέψουν καθ' την ε, ανάπτυξη αυτής της πολιτικής, να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να παραμείνει εν ζωή ο κλάδος αυτός. Νομίζω λοιπόν πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να στηρίξει αυτή την τάση στήριξης θέσεων εργασίας και στην τελική ψηφοφορία εμείς δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να σας στηρίξουμε ε, γιατί η πολιτική μας είναι αυτή. Ευχαριστώ, Ντάμπορ Σκρέτς. Μόλις κατέφτασε, άρτη αφηχθείς ακριβώς, να ε, πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που καθυστέρησα. Είχα μια ανελημμένη υποχρέωση. Αλλά ε, πρόλαβα. Λίγα λόγια κι εγώ. Για την έκθεση του κυρίου Τέλετσκα. Η δουλειά που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ απαιτητική. Και η απόδειξη είναι ότι η ψηφοφορία θα καθυστερήσει στην Επιτροπή μας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει συνταχθεί για να μειωθούν και οι εκπομπές του κλάδου της αεροπλοείας. Πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν να δώσουμε τη σωστή κατεύθυνση με τις τροπολογίες μας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εν μέρη μπορώ να στηρίξω όσα συζητήσαμε και συμφωνήσαμε στις συναντήσεις των σπιωδών. Υπάρχει όμως ένα πράγμα το οποίο ε, δεν με βρίσκει σύμφωνο γιατί δεν ξέρω αν είναι μια σωστή στατηγική επιλογή. Όλος ο τομέας της αεροπλοίας δεν μπορεί να να εξετάζεται και να αντιμετωπίζεται μόνο από την οπτική γωνία της ε, κερδοφορίας. Ασχέτως των διεθνών προτύπων και της συμφωνίας της ΕΚΑΟ για τη μείωση των εκπομπών, ασχέτως ότι αυτό μας ε, βρίσκει σύμφωνους, ας προσπαθήσουμε να στηρίξουμε την έρευνα και την ανάπτυξη. Όχι μόνο στο έδαφος, αλλά και στα αεροσκάφη. Δηλαδή να παράγονται λιγότερες εκπομπές. Να αναφέρω απλώς ότι το άλλο θέμα που απασχολεί την Επιτροπή μας είναι ο τουρισμός και η Ευρώπη θέλει να είναι τουριστικός προορισμός. Αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι θα έρχονται και μάλλον με αεροπλάνο. Σε ό,τι αφορά τις ε, εκπομπές, 45% των εκπομπών των εκπομπών που πρέπει να περιορίσουμε ε, προέρχονται από τον κλάδο της αεροπλοείας. Κάτι που λοιπόν που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. ένα ακόμα στοιχείο που μας ανησυχεί με κάποιες από τις ε, συμβολές της συνεισφορές μας διαταράσσουμε κάπως τις σχέσεις καλές συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών φορέων των διαφορών κρατών μελών οι οποίοι προσπαθούν να μειώσουν τις εκπομπές μέσω των καυσίμων. Σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορώ να συμφωνήσω με την διατροπικότητα στον ευρωπαϊκό ουρανό. Αυτή είναι μια ιδέα που ακόμη δεν έχει οριστεί σαφώς. Οπότε καλό θα ήταν να βασιστούμε σε παγιωμένες καλές πρακτικές ή σε αυτές που έχουν προκύψει προκειμένου να περιοριστούν οι εκπομπές. Αυτό που προέχει είναι να προστατεύσουμε τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και τα δικαιώματα των επιβατών. Να επιμείνω επίσης τους ανθρώπους με περιορισμένη κινητικότητα, με αναπηρίες. Στην διατροπική αυτή ε, αντιμετώπιση των συγκοινωνιών, των μεταφορών, θα πρέπει να προβλέψουμε τη δυνατότητα και σε ανθρώπους που θέλουν να πάρουν το αεροσκάφος να μπορούν να επιλέξουν μεταξύ και άλλων τρόπων μεταφοράς. Είναι πολύ σημαντική αυτή η τροπική μετατόπιση, για να την πω έτσι. Ε, θα το ε, επισημάνω αυτό και στι τροπολόγίε. Με ευχαριστώ τον κύριο Τερίτσκα για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και νομίζω ότι στις μελλοντικέ μα συνεδριάσεις θα ε, καταλήξουμε σε ένα ικανοποιητικό για όλου αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κόχ, θα ήθελα να πω στους διερμηνείς ότι συνεννοηθήκαμε η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού φράζεται στα γερμανικά φεκέρ και τουρισμού. ο τουρισμό και όχι φεκέρ, που είναι ένα συνώνυμο στα γερμανικά. Αυτό αφορούσε τη γερμανική καμπίνα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και τον Μπάβελ Τέλετσκα για τις εξαιρετικές ε, συμβιβαστικέ προτάσεις του. Τρία μικρά σχόλια για τη συμβαστική πρόταση δύο είναι καλύτερο να τονίζουμε την ε, ε, εφαρμογή και υλοποίηση των μέτρων που αφορούν τον ευρωπαϊκό ουρανό για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, στο συμβιβασμό 23, καλά κάνετε και επιλέγετε μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο. Ε, αλλά μετά από κάθε τρομοκρατική επίθεση ή απόπειρα δεν θα πρέπει αυθόρμητα και θερμό να παίρνουμε κάποια μέτρα, αλλά να έχουμε κάποια πιο συγκροτημένη προσέγγιση. Ε, θέλω να σε πείσω και την προσοχή στην 323 δική μου τροπολογία για το δικό, διτό σύστημα ανάπτυξης και εκπαίδευσης καλύτερα ε, ε, θεωρία και πράξη. Δεν αρκεί μόνο το πανεπιστήμιο αλλά θα πρέπει να έχουν και επαφή με την αγορά οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον κλάδο. Ιδιαίτερα όπως είναι η αεροπορία που είναι πάρα πολύ διεθνής οι μεταφορές και διεθνές στο επίπεδο εργασίας. Ε, και ως μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης χαίρομαι που η γνωμοδότηση της Αρμόδιας Επιτροπής ε, λήφθη υπόψη για τα εργασιακά και τα γενικότερα συνθήκες εργασίας. Ευχαριστώ πολύ και τώρα η Γκεζίνε Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ τον Παύλ Τέλιτσκα. Έχουν υποθεί τα περισσότερα, είναι πολύ καλή έκθεση, πολύ ισόρροπη και παρόλο που είναι σχετικά περιορισμένη σε έκταση, αναφέρεται σε πολλά θέματα. Να σας πω εγώ δύο πράγματα που με ενδιαφέρουν πολύ. Το ένα που έχει υιοθετηθεί για τα ιδιωτικά αεροσκάφη, τα ε, τζετ, τα ιδιωτικά, γιατί όταν μιλάμε για αεροπορία σκεφτόμαστε όλοι τις μεγάλες ε, εταιρείε ε, αερομεταφορών, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις μικρότερες και στα αεροδρόμια και να βλέπουμε ποιος μπορεί να προσφέρει ποιες υπηρεσίες και ποιος όχι. Τώρα, το δεύτερο για τους λεγόμενους αυτούς αυτονικοδρόμους των εθέρων, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, η Νέσα για άλλα... Τρελό ακούγεται. Τι είναι αυτό, αυτοκινητόδρομοι στους εθέρους. Δεν είναι τρελή ιδέα γιατί θα αυξηθεί η κίνηση ε, στους εθέρες. Κοιτάξτε στην Ευρώπη αυτό το ζιγζάκ που γίνεται. Αυτό είναι ο στόχος του ευρωπαϊκού ουρανού, να έχουμε περισσότερη κίνηση και στον αέρα. Δεν είναι κακιά ιδέα Μπορεί να φαίνεται τρελό εκ πρώτη όψεω και από τη διατύπωση τώρα τι είναι αυτό αυτοκινητόδρομη στον αέρα, αλλά πάση περιπτώσει ξέρουμε τι λέμε και περί τίνο πρόκειται. Και αφορά γενικά ε, το σύνολο ε, του κλάδου και το μέλλον του κλάδου. Ευχαριστώ, Ιζαμπέλα Δεμόντε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω ε, τον εισηγητή, τους και εισηγητές, για τη δουλειά που έχουν κάνει και για τους συμβιβασμούς. Ε, θα ήθελα να πω κάτι για τα περιφερειακά αεροδρόμια, γιατί έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν και για την αποσυμφόρηση των βασικών αερολιμένων, αλλά και για μια τοπική ανάπτυξη που είναι πολύ σημαντική και για τον τουρισμό. Άρα λοιπόν Ε, μπορεί να θεωρείται ότι δεν έχει ιδιαίτερε επιπτώσει για τα κράτη-μέλη, αλλά έχει σημασία. Και επίση έχει σημασία να επιμείνουμε στη διάσταση της ευελιξίας ε, και της ελαστικότητας. Όταν ένας τοπικός ε, φορέας χρειάζεται μια υπηρεσία, ε, χρειάζεται να υποβάλει υποψηφιότητα, αίτηση κτλ. για ενίσχυση για τις επενδύσεις αλλά και για τη λειτουργία. Στην ε, συμβαστική 20 είναι θετικό ότι δόθηκε ιδιαίτερη αξία στα duty free που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, βιωσιμότητα, την οικονομική βιωσιμότητα των αεροδρομίων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ξαναζήτησε το λόγο η ευχαριστω πολυ μονο Μάισνερ. Γιατί πρέπει να πω στον υφιστάμενο κανονισμό, λέει πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ξεπεράσουμε τις περιφερειακές ε, συμφορήσεις, δηλαδή την περιφερειακή συμφόρηση Regional Bottleneck. Οπότε, στην τεχνολογία που έχουμε στη νέα πρόταση, σύμφωνα με τα όσα λέει ο συγητής, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε πως μπορούμε με τον τρόπο αυτό να ξεπεράσουμε καταστάσεις, για παράδειγμα, νόμιμης απεργίας. Δηλαδή, μιλάμε για βιομηχανικέ σχέσει ουσιαστικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάποιε περιπτώσει τεχνολογίε αυτέ για αυτό το οποίο ε, ονομάζει Commission Regional Bottlenecks. Βέβαια, ίσως θα πρέπει να μα ξεκαθαρίσουν ακριβώ περί τίνο πρόκειται, γιατί αυτή είναι η βασική ε, διαφορά για μένα, γιατί σήμερα η διατύπωση συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα, εάν θέλαμε να χρησιμοποιηθεί, γι' αυτό να γίνεται. Ευχαριστώ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Φίλιπ Κονέλης από την Γενική Διεύθυνση MOVE. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση την οποία προετοίμασε και η οποία νομίζω ότι σε γενικές γραμμές στηρίζει τη δική μας ε, στρατηγική για την αεροπλοεία. Και να σας πω πως καλωσορίζω το γεγονός πως στηρίζεται τόσο πολύ από την Επιτροπή σας η έκθεσή του, γιατί νομίζω ότι είναι μάλλον εκ μέρους όλων των πλευρών. Και αυτό για μας είναι θετικό, μια και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε με τη στρατηγική μας και να την εφαρμόσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Λοιπόν, για δύο σημεία τα οποία ε, έχουν ε, ακουστεί για τη συζήτηση και για τις τροπολογίες παρόλο που δεν έχουμε δει ακόμα τους συμβιβασμούς για την εξωτερική πολιτική αεροπλοείας και για την περιφερειακή διασυνδεδημότητα. Σημότητα. Για την εξωτερική πολιτική να σας πω πως αυτή τη στιγμή προχωράμε ταχύτατα. Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με αρκετέ τρίτες χώρες επί τη βάση της εντολής που λάβαμε, τον Ιούνιο μάλιστα. Και ο θεμητός ανταγωνισμός είναι κομμάτι αυτών των συζητήσεων που διεξάγουμε. Δεύτερον, για τα εξωτερικά μας θέματα με ιδιαίτερη επιμέλεια ασχολούμαστε με μια πρόταση η οποία θα αντικαταστήσει τον 868 κανονισμό και στόχος μας είναι και ελπίδα μας να μπορέσουμε να τα καταθέσουμε τα νέα κείμενα το συντομότερο δυνατόν μετά το νέο έτος. Για την περιφερειακή διασυνδεσιμότητα να σας πω πως ε, καταρχήν και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε την ε, διασυνδεσιμότητα εξαιρετικά σημαντική, εξαιρετικά σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλές περιοχές, για παράδειγμα για τις υπερπόντιες ή πολύ απομονωμένες περιοχές που διαφορετικά δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν εύκολα. Υπάρχει λοιπόν μια θετική τάση στην ίδια την ε, βιομηχανία του κλάδου, μια και αυτή τη στιγμή δίδεται μικρότερη σημασία για ταξίδια μέσω κόμβων, αλλά περισσότερη σημασία για ταξίδια που συνδέουν απευθεία αυτά τα οποία θα ε, χαρακτηρίζαμε δευτερεύοντα αεροδρόμια. Τώρα, για το δυναμικό, για τα περιφερειακά αεροδρόμια, πιστεύουν πως θα πρέπει να έχουν το δυναμικό για να ανταποκριθούν στη ζήτηση. Αλλά το δυναμικό αυτό θα πρέπει να είναι το κατάλληλο. Ούτε υπερβολικά πολύ, ούτε υπερβολικά λίγο. Δεν θέλουμε βέβαια να έχουμε άδεια αεροδρόμια, ούτε όμως να μην υπάρχουν εκεί που χρειάζονται. Υπάρχουν τα εργαλεία αυτή τη στιγμή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Το κάνουμε ήδη, έχουμε και τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις, έχουμε το ΕΦΣΙ και την ε, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω αυτού και όλους τους κανονισμούς που θα μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε την περιφερειακή διασυνδεσιμότητα. Τέλος κύριε Πρόεδρε για τον ε, ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό να σας πω πως και εμείς και εμείς πραγματικά είμαστε εκνευρισμένοι από την έλλειψη προόδου σε αυτή την πρόταση ε, λόγω της διαφοράς που υπάρχει μεταξύ κρατών για το Γεβραλτάρ. Χαιρόμαστε για κάθε στήριξη μας προς το κοινοβούλιο εκεί και για τους αυτοκινητοδρόμους των εθέρων. Θα το σκεφτούμε Βέβαια όταν λέμε αυτοκινητόδρομοι συνήθως σκεφτόμαστε κίνηση, θόρυβος, καυσαέρια. Ε, είναι μάλλον το αντίθετο αυτό που πρέπει να πετύχουμε στους ουρανούς και καλό θα ήταν να έχουμε μια ελεύθερη ροή στον αέρα έτσι ώστε να, υπάρχουν η δυνατότητα, να υπάρχει δυνατότητα να πετάνε απευθείας ακολουθώντας ε, μια ευθεία πορεία τα αεροπλάνα χωρίς να χρειάζεται να κάνουν παρακάμψεις παρόλο που σε κάποιες περιοχές μπορεί να υπάρχουν ε, προβλήματα που σήμερα οδηγούν σε τεράστιες παρακάμψεις που δεν εξυπηρετούν ούτε τον επιβάτη που κάθεται για περισσότερες ώρες στο αεροπλάνο ούτε και τις εταιρείε. Θα το σκεφτούμε να δούμε τι θα προκύψει από την έκθεσή σας και σας ευχαριστώ και πάλι για την γενικότερη στήριξη που μας προσφέρετε. Ευχαριστώ πολύ. Πάλι ο ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να αντιδράσω σε κάποια από τα σημεία που έθιξαν οι συνάδελφοι. Για άλλη μια φορά, εκτιμώ τα σχόλιά τους. Όπως είπαν και οι σκιώδεις από την αρχή, είναι πολύ καλή η ατμόσφαιρα και είναι πολύ καλό το επίπεδο συνεργασίας μας. Μερικές παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, για την έννοια των αυτοκινητοδρόμων του ουρανού. Ναι, όπως είπε και η Επιτροπή, εδώ θέλουμε ελεύθερες συγκοινωνίες. Και δεν θέλουμε στα στρατηγική να υπάρξουν υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες. Απλώς η ουσία είναι να συνεννοηθούμε εμείς ως σκιώδεις για αυτή την έννοια. Το είπε και η κυρία Γιάλα Σέντερ. Δεν θα πρέπει τα συνταγματικά και άλλα δικαιώματα των εργαζομένων να φυγούν. Το δικαίωμα στην απεργία και το, το καθεξής. Είχατε διασφάλιση την ε, εγγύηση ότι δεν θα παραβιαστούν αυτά τα δικαιώματα με τι διατάξει που προτείνονται. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε. Να συζητήσουμε την ε, ε, έννοια αυτή των λεωφόρων του ουρανού. Αλλά στην ουσία θέλουμε να επιτρέψουμε την ελεύθερη ροή των ε, αερομεταφορών με τη μεγαλύτερη δυνατή με το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό διασύνδεσης. Πάντως, εάν χρησιμοποιεί χρησιμοποιηθεί ο όρος διακοπή, διαταραχή, δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση την απεργία. Εννοούμε κάτι που να μην μπλοκάρει την ελεύθερη ροή όπως σεισμοί και φυσικά φαινόμενα. Ε, πρέπει να διευκρινιστεί αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο να πω επίσης ότι Και ίσω επειδή η κυρία Κούνα δεν μπορούσε να... Κλούνε δεν μπορούσε να είναι εδώ χθε, θα τα δούμε με Mm. Νομίζω ότι η μέρημνα αυτή μπορεί να καλυφθεί και να καταλήξουμε σε κάποια μορφή συνεννόηση, όπως είπα. Θα βασιστούμε και σε όσα υπάρχουν και όσα θα μπορούσαν να, να υλοποιούνται καλύτερα. Έχουμε συγκεκριμένου στόχου και ο σκοπό είναι να πάμε στο δυνατόν μακρύτερα για τι κοινωνικέ πτυχέ. Αυτό το έθεσαν αρκετοί συνάδελφοι, αλλά ελπίζω να συμφωνούν ότι στην πρόταση των ξεμεμπαστικών τροπολογιών τα ζητήματα αυτά καλύπτονταν. Το θέμα είναι να συζητήσουμε τι βαθμό λεπτομέρεια θέλουμε. Όπω είπα από την αρχή, αυτή είναι μια στρατηγική για την αεροπλοεία που θέλει να υπογραμμίσει ζητήματα που μπορεί να μην έχουν άμεση σχέση με τις μεταφορές, έχουν, ε, είναι σκόπιμο να αναφερθούν, αλλά δεν θέλουμε να τα εξηγήσουμε σε λεπτομέρειες για την δική μας αρμοδιότητας. Και θα φροντίσουμε στην τελευταία συνεδρίαση των ε, σχεδόν να δώσουμε μια καλύτερη προβολή στο κείμενο, στα κοινωνικά ζητήματα τώρα για, το, για τη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι είναι σαφές το κείμενο. Η έκθεση δηλαδή. Ε, με τον 868 έχουμε συγκεκριμένε απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά υπάρχουν και διμερεί συμφωνίε που προκύπτει από την έννοια ιδέα πρόταση του δικαίου, του δικαίου ανταγωνισμού και της σχετικής ρήτρας. Θα επιμείνουμε σε αυτό, καθώς συμφωνία υπάρχει και να πω και στους συναδέλφους σοσιαλιστές και δημοκράτες ότι το περιδικαίου θέμα για τις κρατήσεις, τα εισιτήρια και το καθεξής βεβαίως θα ληφθεί υπόψη. Και έπειτα για τις ε, περιοχές, τα αεροδρόμια που βρισκόνται σε περιφερειακότερες θα πρέπει να έχουμε μια σωστή ισορροπία. Αυτό που είχα βέβαια εγώ υπόψη είναι η πυκνοκατοικημένες περιοχές όπου έχουμε πολλά αεροδρόμια που δεν λειτουργούν επαρκώς και χάνουμε μεγάλες δυνατότητες κερδοφορίας. Εδώ ε, ο συνδυασμός των τρόπων συγκοινωνιών έχει μεγάλη σημασία. Στις περιοχές αυτές δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος μεταφοράς, ούτε θα πρέπει να μελήσουμε τα αεροδρόμια αυτά. επειδή δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη η κερδοφορία τους. Αναφέρθηκε το Γιβραλτάρ, αλλά δεν αναφέρεται αυτολεξή στο κείμενο. Το τι μπλοκάρεται στο Συμβούλιο σε σχέση με τόσα προτείναμε είναι πράγματα για τα οποία εμείς μεταξύ μας συμφωνούμε. Να είναι ξεκάθαρο. Και ε, χαίρομαι που συμφωνούμε. Και μια από τις τελευταίες μου παρατηρήσεις Λυπάμαι που δεν είναι εδώ ακόμη η κυρία Κονέτσινα. Ίσως επειδή δεν ήταν στη συνεδρία των σχεδόν. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις. Αλλά το θέμα που έθιξε υπάρχει στο κείμενο. Με τη λογική που ανέπτυξα. Ελπίζω ότι θα το ξαναδούμε, αλλά δεν ανάγκη να πούμε τώρα τα πάντα γι' αυτό και για την ΙΚΑΟ. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι συνάδελφοι, κάποιοι από εμά, θα δέχονταν όσα λέει η ΙΚΑΟ. Ίσως έχει πάει ε, ίσως θα μπορούσε να έχει πάει πιο μακριά, αλλά αυτό που έχουμε από την ΙΚΑΟ είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Σε αυτό που να βασιστούμε για το μέλλον. Α ε, επιδιώξουμε να έχουμε διατύπωση στο κείμενο, όπω τώρα έχουμε, που να είναι αρκετά σταθερή. Ένα καλό συμβιβασμό δηλαδή. Συνολικά, πρόεδρε και συνάδελφοι, αυτά έχω να πω. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος των ανησυχιών που ακούστηκαν ως προς το σχεδιασμό της στρατηγικής μας αντικατοπτρίστηκαν στο βαθμό που ακολουθήσαμε την προσέγγιση την οποία είχαμε συμφωνήσει στην αρχή της διαδικασίας. Το είπαν και οι συνάδελφοι και επιβεβαιώθηκε. Νομίζω ότι σε λίγες μέρες, δέκα μέρες το πολύ, θα έχουμε τα τελευταία συνεδρία των Σκιωδών και θα είμαστε στην ώρα μας για την ψηφοφορία στις 5 Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε λοιπόν, 5 Δεκεμβρίου ψηφίζουμε. Πάμε στο επόμενο θέμα. Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοεία. Η συγγήτρια είναι η κυρία Γκεζίνη Μάισνερ, η οποία έχει το λόγο αμέσω. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πάμε λοιπόν από τον αέρα το νερό στην εσωτερική ναυσιπλοεία, ποτάμια, κανάλια κτλ. Αυτό ο κόσμος δεν το ξέρει παντού στην Ευρώπη, δεν αφορά όλα τα κράτη-μέλη, δεν έχουν εσωτερική ναυσιπλοεία όλοι, παρόλα αυτά είναι σημαντικό το θέμα. Και καλό είναι να κοιτάξουμε πώς θα προετοιμάσουμε, ε, προετοιμάσουμε συγγνώμη, το μέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης ηγητές. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητική συνεργασία. Ο πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια. Κάνετε πολύ φασαρία. Το λόγο έχει και Σίνε ναι, Μάισνερ. Ναι, όταν μιλάς για ποτάμια, μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, συνεχίζω. Ε, σε ευχαριστίες ήμουνα ε, τους Κιώδης και τους, ε, την πολιτική σύμβουλο Ντομινίκ από τη Γραμματεία, γιατί την έψαχνα εδώ μπροστά κάθεται. 252 είναι οι τροπολογίες, 23 οι συμβαστικές. Οι περισσότερες τροπολογίες έχουν ληφθεί υπόψη στις συμβαστικές. Βεβαίως δεν κέρδισαν οι πάντες, ούτε καν εγώ ως εισηγήτρια. Ο καθένας έπρεπε να βάλει λίγο νερό στο κρασί του και να υποχωρήσει δύο σκιώδεις, μάλλον δύο συνεδριάσεις σχεδόν εισηγητών χρειάστηκαν. Χτες ήταν η δεύτερη και τελειώσαμε και μισή ώρα νωρίτερα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν δυνατότητες και τα πήγαμε καλά στη συνεννόηση. Να πω λίγο σύντομα στο περιεχόμενο. Ποιο είναι ο στόχο και παραμένει γιατί δεν έχει τελειώσει, να υπάρχει εναρμονισμένη εκπαίδευση και κατάρτιση για την εσωτερική νευσιπλοεία στην Ευρώπη. Γεια σου, Πέτερ Βαντάλεν. Ε, τα ξέρει πολύ καλά αυτά ο κύριο Βαντάλεν. Ε, εσωτερική ναυσιπλοεία στην Ευρώπη δεν ήταν εναρμονισμένη. Μιλώ πάντα για την επαγγελματική κατάρτιση. Χρειάζεται οπωσδήποτε γιατί ε, λείπει ε, δυναμικό και άνδρες και γυναίκες και το τονίζω γιατί και οι γυναίκες ξέρουν ε, τέτοια επαγγέλματα ε, και για να υπάρξει κινητικότητα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση. Το ε, πιο δύσκολο ήταν το πεδίο εφαρμογής και εξαιρέσεις σε αυτή την υπόθεση. Ξέρω ε, ότι δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι με αυτό στο οποίο καταλήξαμε. Υπάρχουν χώρες όπως είναι η Μάλτα. Η Μάλτα εκπαιδεύει ναυτικούς χωρίς να έχει ποτάμια. Εκπαιδεύει προφανώς ναυτικούς για τη θάλασσα και δεν μπορεί να εξαιρεθεί. Η Φιλανδία ε, έχει πολλές λίμνες που δεν συνδέονται με την υπόλοιπη Ευρώπη και για να ε, ε, αρμενίζεις τη λίμνη χρειάζεσαι άλλα προσόντα από το να είσαι σε ένα ποτάμι με ένα ποταμόπλιο. μετά, άλλα θέματα είναι ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι να γνωρίζει κανείς ε, τα ποτάμια. Τα ποτάμια και οι διαδρομές έχουν την ιδιαιτερότητά τους. Ε, στη Γερμανία έχουμε σωρίνο τη Λορελάη που είναι ένας βράχος περίφημος και το τραγουδάμε και όλες και έχει και θρύλους. Ο Δούναβης έχει τις δυσκολίε και η Γαλλία βλέπω το Ρενό Μιζουλιέ εδώ πέρα έχει ποτάμια ε, που χρειάζεται να γνωρίζει κανείς το ποτάμι για να ταξιδεύει σε αυτό. αυτά. Ε, είχαμε και την πρώτη ευρωπαϊκή Επίτροπή για την είσοδο στο επάγγελμα από άλλα επαγγέλματα και διάφορα άλλα θέματα τεχνικά ε, ε για ναυτόπεδες, ε, ναύτες, ε, κυβερνήτης. Υπάρχει μια επιτροπή που λέγεται ΣΕΣΝΗ που είναι Επιτροπή του Ρήνου και κάποιες άλλες που ρυθμίζουν αυτά τα πράγματα για τη συμπεριφορά ε, ε, στα ποτάμια κατά την εσωτερική ναυσιπλοεία. Υπάρχει και επιτροπή ολόκληρη που λέγεται River Commission. Ε, για το χρονοδιάγραμμα γνωρίζουμε ότι οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες ζήτησαν να μην ψηφίσουμε αύριο αλλά να το αναβάλουμε. Εγώ θα ζητούσα πάρα πολύ να ψηφιστεί αύριο ε, είναι όριμο το θέμα, έχει κυκλοφορήσει κατάλογο ψηφοφορία από τη Δευτέρα. Εχθέ συμφωνήσαμε, ε, ψηφίσουμε σε μεγάλο βαθμό. Βεβαίω θα πρέπει να σκεφτούμε ε, ότι θα πρέπει να είμαστε μεθοδικοί και όχι βιαστικοί. Μα είμαστε μεθοδικοί, μια χαρά τα έχουμε κάνει. Απλώ να σκεφτούμε το εξή. Οι Σλοβάκοι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Πραγματικά έχουν αφαιρεθεί στην νομοθεσία και περιμένουν να αρχίσει ο τριμερή διάλογο. Ισχύει καμιά φορά ε, να βιάζεται πιο πολύ το Συμβούλιο από εμά και να μας περιμένει. Αν αρχίσουμε τώρα τις χρονοτριβές και τις ολιγορίες δεν θα ολοκληρωθεί στον τριμερή διάλογο, αλλά έχει και την επόμενη Προεδρία που είναι η Μάλτα, η οποία βέβαια δεν πολύ ενδιαφέρεται για το θέμα, αλλά φοβάμαι αν δεν κλείσει τώρα στη Σλοβακική Προεδρία θα πάει στις καλένδες. Ε, παρακαλώ λοιπόν να ψηφίσουμε αύριο για να αρχίσει ο τριμερής διάλογος. Ευχαριστώ. Ε, εγώ νομίζω Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ε, χαιρετήσω την εισηγήτρια για την εργασία της πραγματικά με πολύ μεγάλη ε, δεξιοτεχνία το χειρίστηκε το θέμα αυτό. Είναι περίπλοκο, είχαμε λίγο χρόνο, καταλήξαμε σε μια πολύ θετική ε, στάση και θέση και την υποστηρίζω βεβαίως να ψηφίσουμε αύριο έχει ολοκληρωθεί αυτό το θέμα, αυτή η εργασία και είναι γεγονός ότι μας περιμένει το Συμβούλιο. Τώρα, επί της ουσίας, 23 συμβαστικές τροπολογίες μας βρίσκουν σύμφωνους γιατί ε, ακολουθούν τη γραμμή που είχε χαράξει το ΕΛΚ. Ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό για το Βοτάμιο δίκτυο ε, και ε, ε, εξαίρεση για όλα τα ποτάμια που δεν συνδέονται με το δίκτυο. Υπάρχουν εξαιρέσει πάρα πολύ ιδιαίτερε, πάρα πολύ περιορισμένες και τοπικές επαγγελματική κατάρτιση που να μην έχει αποκλεισμού και να δίνει επαγγελματικέ δεξιότητε και προσόντα στους Ευρωπαίους, σταδιακή υιοθέτηση αυτού του συστήματο για να μπορέσει να προσαρμοστεί ο κλάδο και μεγάλη συνεννόηση και σχέση με τις ΕΣΝΗ και τι άλλε επιτροπέ που θα ορίσουν του ε, μελλοντικού κανόνε. Όλα αυτά λοιπόν μα βρίσκουν σύμφωνους. Θα ήθελα όμως να επιμείνω σε ένα σημείο που έχει τη σημασία του και δεν βρήκε τη θέση του στο ε, συμβιβασμό το πεδίο εφαρμογής. Ορισμένοι θεωρούν ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στα κράτη-μέλη που έχουν κέντρα εκπαίδευσης ή και πλωτά ποτάμια. Αυτό μπορεί να φαίνεται λογικό, αλλά ειλικρινά είμαι πεπισμένος ότι η κάθε ευρωπαϊκή νομοθεσία, είτε είναι κανονισμός είτε οδηγία, θα πρέπει να φαινεται λογικο αλλα ειλικρινα ειμαι πεπισμενο οτι η εφαρμογή παντού. Ε, το δικαστήριο ε, αναγνώριση το δικαίωμα στις χώρες που δεν του αφορά να μην μεταφέρουν την οδηγία, αλλά καλό θα ήταν να έχουμε και μια συνοχή και όχι ένα σύνολο εθνικών εξαιρέσεων στην νομοθεσία μας. Αυτά. Ε, γενικότερα δεν μπορώ παρά να εγκρίνω την έκθεση αυτή και να την υποστηρίξω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πέτερ Παντάλεν. Πρόεδρε, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγήτρια ειλικρινά ε, ε, έχει χειριστεί το θέμα πάρα πολύ επαγγελματικά, νυφάλαια και ρεαλιστικά. Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ε, για μένα αυτό που έχει σημασία είναι οι συμβιβαστικέ τροπολογίε για τις επιτροπές των ποταμών. Έχουμε τρεις τέτοιες επιτροπές στην Ευρώπη που θέλουμε να συμμετέχουν περισσότερο για τα επαγγελματικά προσόντα, για την εναρμόνιση και την αναγνώριση. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάρα πολύ ισχνή και δίνει πολύ μικρό χώρο σε αυτέ τις τρεις επιτροπές. Εμεί το έχουμε εξισορροπήσει ε, με τι διάφορε συμβαστικές τροπολογίε. Επίση, συζητήσαμε πολύ ε, τι θα γίνει με την κατάρτιση, τι θα γίνει με την εμπειρία που χρειάζεται στην αυσιπλοεία, πόσους μήνες ε, πρέπει να βάλουμε, πόσα χρόνια. Ε, θα πρέπει να παραμείνουμε, πιστεύω, στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί ε, ξέρουν και λαμβάνουν υπόψη την πρακτική στα κράτη-μέλη για να κάνουν τις προτάσεις αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό έχει εφαρμοστεί και έχει αποδειχθεί στην πράξη δηλαδή και ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και η επαγγελματική κατάρτιση είναι πάρα πολύ ψηλής ποιότητας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ ισορροπημένες αυτές οι συμβαστικές τροπολογίες, τις υποστηρίζουμε σχεδόν όλες, μία ή δύο όχι, το τελικό αποτέλεσμα οπωσδήποτε και το χρονοδιάγραμμα που προτείνει η συγκήτρια ε, μας βρίσκει σύμφωνους επίσης να ψηφίσουμε αύριο και μάλιστα να το βάλουμε και πρώτο θέμα στη μέση διάταξη αν με ρωτάτε. Ευχαριστώ. Η Κλαούντια Ταπαρντέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την συμμετοχή του και τη σκληρή του δουλειά. Η έκθεση για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσώπων στην εσωτερική νοσηπλοεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, διότι θα συμβάλλει στην πρόθεση τη κινητικότητα αυτών τον τομέα, αλλά είναι και ένα θέμα αρκετά περίπλοκο, διότι χρειάστηκε να μπούμε σε πολλέ λεπτομέρειε. Είναι πολύ τεχνικό Επίσης, θέλω να πω ότι κάποιες φορές οι απόψεις των συναδέλφων, όπως αντικατοπτρίζονται τι τροπολογίε, αποκλίνουν μεταξύ τους και αυτό φαίνεται και στο κείμενο που έχετε μπροστά σας. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, η ομάδα μας δεν θα στηρίξει τις τροπολογίες που προβλέπουν εξαιρέσεις, παρεκκλήσεις, διότι αυτό θα παραβίαζε και θα ερχόταν σε αντίφαση, θα αντίκειτο με το ίδιο το πεδίο της οδηγίας. Αυτό που θέλουμε είναι ένα σύστημα συνεκτικό, συνεπές, που να μπορεί να εφαρμοστεί ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη-μέλη και να επιτρέψει σε οποιονδήποτε πολίτη το επιθυμεί να ε, εργαστεί από τον επαγγελματικό κλάδο. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι το θέμα αυτό αγγίζει τις αρμοδιότητες και άλλων ε, επιτροπών στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι όλες οι επιτροπές που ασχολούνται με την ε, καλή κατάσταση διαφόρων ποταμών ανά την Ευρώπη και όλες οι ενώσεις πολιτών ε, βλέπουν να τους καλύπτει και να τους προστατεύει αυτή η οδηγία. Θέλουμε να έχουμε σαφή πρότυπα ως προς την ε, επίβλεψη της υλοποίησης αυτής της οδηγίας και ελπίζουμε ότι κάτι τέτοιο ήδη προβλέπεται. Δεν θέλουμε να επιτρέψουμε σε ένα κατομέλο ή ένα άλλο, στο ένα ή στο άλλο κατομέλος ή στην την άλλη επιτροπή να επιβάλλουν μέτρα περιοριστικά. Γι' αυτό θα συναντηθούμε ξανά ε, σε επίπεδο σκιωτών εισηγητών για να καταλήξουμε σε μια τελική θέση για όλες τις συμβαστικές τροπολογίες. Επίσης, θα ήθελα να ζητήσω από την Κιεζίνε κάποιες λεπτομέρειες για την τροπολογία 54. Προς στιγμή δεν είμαι βεβαία ότι οι αλλαγές που προτείνονται είναι υποφελής. Ποια ήταν η συλλογιστική για τις προτάσεις που γίνονται στην ε, τροπολογία 54. Διότι ένα από τα πράγματα που είπαν πολλές ε, φορές οι ενδιαφερόμενοι στις διαβουλεύσεις που είχαμε είναι ότι συχνά οι εργαζόμενοι προέρχονται από χώρες που δεν έχουν εσωτερικούς δρόμους ναυσιπλοείας. Οπότε δεν υπόκεινται σε όσο προβλέπει αυτή η οδηγία. Θα πρέπει λοιπόν η τροπολογία 54 να διευκρινιστεί. Ευχαριστώ. Η Μέρη Κριστίνα Γνώτσου. Δεν θέλω το λόγο, λέει κύριε Γνώτσου. Καλά, είναι σε άλλα τότε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω οι ε, εισηγητέ και σκιώδεις εισηγητέ και να σας πω πως αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς συμπεριλήφθηκαν δύο στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την δημιουργία αυτού του ευρωπαϊκού ε, καθεστώτος, για να το πω έτσι, ε, ε, με αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι η μόνη, η οποία έχει βέβαια την εμπειρία, αλλά για τα ποτάμια πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και κάποιες καινούργιες ιδέες και να σας πω πως για την τροπολογία 176 η εισηγήτρια την έλαβε υπόψη, εντάξει, και μετά ρωτώ την εισηγήτρια και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 125 που προτείνουμε στην Κομισιόν να παρουσιάσει ένα νομικό πλαίσιο για αυτόν το ταχυγράφο που θα χρησιμοποιούν ε, στα πλοία, στα ποτάμια, που είναι μια ιδέα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τουλάχιστον για όσους ε, φέρουν επιβάτες και εμπορεύματα. Λοιπόν, αυτός ο ταχογράφος μας δίνει τη δυνατότητα να καταγράφουμε ακριβώς πώς γίνονται αυτές οι μεταφορές και τι σημαίνει αυτό για την εργασιακή ε, ηρεμία όσων εκεί εργάζονται. Οπότε θα θέλαμε να το δούμε ένα νομικό πλαίσιο που να διέπει ακριβώ αυτέ τι διατάξει. Τώρα πάντα κάμπ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Μάισνερ και τους χειώδεις εισηγητέ. και ήταν περίπλοκη αυτή η υπόθεση, το λέω ειλικρινά. Κοιτάω και τον κύριο Βαντάνερ γιατί τρόμαξα και ο ίδιος. Τι χρειάζεται να μελετήσει κανείς για να ε, κάνει μια οδηγία για πιο ομοιόμορφη κατάρτιση και επαγγελματικά προσόντα στην εσωτερική ναυσιπλοεία. Πρέπει να σας πω ότι το είχα υποτιμήσει το θέμα και έλεγα έλα μωρέ σιγά ένα απλό θέμα είναι να το δώσουμε στην Κεζίνε θα το διεκπαιρεώσει μια χαρά και γρήγορα. Καθόλου. και με τον κύριο Μπιζολιέ που είναι ο σκιώδης ηγητής μας το συζήτησα και πρέπει να σας πω ότι είχαν πολλά τα προβλήματα για την εσωτερική αγορά. Λοιπόν, τώρα το φέραμε αυτό σε ένα αίσιο πέρας και αύριο μπορούμε να ψηφίσουμε. Ακούω από τον κλάδο, αν και δεν είμαι ειδικό ε, καθόλου, ότι υπάρχουν ε, κλάδοι ε, στην ε, εσωτερική ναυσιπλοεία όπου δεν υπάρχει ημερολόγιο καταστρώματος. Υπάρχει κάποια μεταβατική περίοδος για να επιβληθεί αυτό σε κάποια κράτη-μέλη. Και 20 χρόνια θέλουν να βάλουν μεταβατική περίοδο. Πάρα πολλά δεν είναι, μια 20 ετία. Και εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος το λέω αυτό. Μπορεί να μας απαντήσει η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν να απαντήσει η κυρία Μάισνερ, θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την κυρία Τανιέλα Ράσκα. Uh, uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια κυρία Μάισνερ και τους Κιώδης και καταρχάς να πω σε όλους γιατί προβλέφθηκε αυτή η πρωτοβουλία. Εσωτερική ναυσιπλόγια, εσωτερική δρόμη ναυσιπλογίας. Βιώσιμος τρόπος μεταφοράς, φιλικός προς το κλίμα, με δυνατότητα, με πολλές δυνατότητες που τώρα δεν έχουν να χρησιμοποιηθεί, αξιοποιηθεί μάλλον, και με πολλά εμπόδια στην ανάπτυξή του. μέσος όρος ηλικίας 50 ε, ετών στους εργαζομένους, ε, έλλειψη ισορροπίας στην προσφορά των υπηρεσιών στις διάφορες περιοχές, επαγγελματικά προσόντα που χρειάζονται πολύ και ε, η, εργα... η κινητικότητα του... της εργατικής δύναμης είναι κάτι σημαντικό, αλλά και το να διατηρήσουμε το κατάλληλο επίπεδο προστασίας. Πολύ σημαντικό λοιπόν να παραμείνει και η εσωτερική ναυσιπλοεία μέρος της προσπάθειάς μας ε, να είναι διατροπική η διασύνδεση των τρόπων μεταφοράς. Εδώ λοιπόν προκειμένου να είμαστε συνεπείς με τους στόχους μας και συνεκτικοί στην προσέγγισή μας, εξετάζουμε τις διαφορετικές τροπολογίες, διότι δεν θέλουμε να υπάρξει περιορισμός της κινητικότητας των εργαζομένων και η ελκυστικότητα του τομέα αυτού που είναι ο απότερο στόχος της δικής μας της πρότασης. Αλλά να διατηρήσουμε επίσης και το κατάλληλο πλαίσιο νομικής βεβαιότητας και ασφάλειας που μας αφορά και επίσης θα δώσω σύντομα το λόγο και στον συναδέλφο Μάρκ Βάντερ για να εξηγήσει πολύ ε, γρήγορα κάποια από τα σημεία αυτά. Ευχαριστώ κύριε Γκυζίνε Μάισνερ. Er Μα έλεγε ότι θα δώσει το λόγο στον Μάρκο Van Α, καλά. Yes, uh, thank you and uh, also from my... Σας ευχαριστώ και εγώ από πλευράς μου να σας καλημερίσω. Όλους και όλες. Οι ανησυχίε μας έχουν να κάνουν όλο ιδιαίτερως με την δυνατότητα όλοι οι βαθμοί πέραν των, ε, των κυβερνητών να έχουν ε, το σύστημα έγκρισης των δεξιοτήτων. Το σύστημα που έχουμε όμως τώρα είναι απερχαιωμένο. Βασίζεται μόνο στην εμπειρία, ε, τουλάχιστον το νέο σύστημα. Με αυτές τις τροπολογίες το παλιό σύστημα θα συνυπάρχει με το καινούριο, που θα βασίζεται στο κατά πόσο κάποιος έχει τις δεξιότητες που πρέπει όχι. Αυτό θα ακυρώσει τελείως τη δική μας προσέγγιση για την νέα οδηγία. Δεύτερη και βασική μέρημνα, η τροπολογία περιθμών 14. Και εδώ ανησυχούμε. Διότι κάποιοι κίνδυνοι γίνονται λίγο πιο γενικευμένοι, όπω το κριτήριο του υψηλή συχνότητα ατυχημάτων. Αδύνατον για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπιστώσει. Και πολύ δύσκολο να τεθεί σε εφαρμογή. Το ίδιο και η απέτηση σε αυτέ τι διαδρομέ να εκτελούνται πάντοτε ταξίδια. Αυτό ορίζει και επηρεάζει την κυριωτικότητα των εργαζομένων. Επίσης, ο αποκλεισμός προσώπων, ατόμων, από τον χειρισμό περιορισμένων διαδρομών σε λίμνες, όπως αναφέρει η τροπολογία 1, ε, εδώ η συγγήτρια είπε ότι η Φιλανδία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει την εθνική της νομοθεσία. Και πέραν αυτού του ε, θα πρέπει να προβλέψουμε κάτι για τις χώρες ε, όταν δεν καλύπτονται από τη σημερινή νομοθεσία. Αυτό θέλαμε να πετύχουμε με αυτή την πρόταση. Επίσης, ανησυχούμε με την, ε, με την οποιαδήποτε μνήμα σε τεχνικές οδηγίες που έχουν τελείως διαφορετικούς στόχους σε σχέση με αυτήν την οδηγία και σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των προσώπων. Επίσης, η τροπολογία που φύγει την αναγνώριση των ε, πιστοποιητικών ε, των διαφορών χωρών, των εθνικών πιστοποιητικών, θα πρέπει να συμμορφούνται και με τα πρότυπα και τι προδιαγραφέ τη Συμφωνία ΓΚΑΤ. Και αυτό δεν αντικατοπτρίζεται αυτή τη στιγμή στο κείμενο, όπω με την τροπολογία 4 Επιφυλασσόμαστε λοιπόν ω προ τη θέση μα για τι ε, συμβαστικέ τροπολογίε, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλουμε να έχουμε επικοδομητική συζήτηση και συνεννόηση μαζί σα για να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ και πάλι τους, ε, τον, την εισηγήτρια και του κοιόδη εισηγητέ για την πολύ στενή του συνεργασία μαζί μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα την Ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις αντιδράσεις. Σας είπα, δεν μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε τους πάντες, ούτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κάναμε ευτυχισμένη απολύτως. Ε, τι να κάνουμε, έχουμε κάποιες ιδέες στο Κοινοβούλιο και όταν έχουμε θέση στο Κοινοβουλίο, είναι θέση του Κοινοβουλίου. Και μπαίνουν και κάποιες εμπειρίες κάποιων κρατών μελών και στην εσωτερική ναυσιπλοεία πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο πολύ διαφορετικά τα ποτάμια και τα κανάλια, είναι πολύ διαφορετικές και οι παραδόσεις και οι κουλτούρες και οι εμπειρίες και το είπε και η Κλάουντια, ε, ε, έχουμε κάνει διαφορετικές τροπολογίες και μάλιστα από την ίδια πολιτική ομάδα. Εγώ προσπάθησα να κάνω ένα συμβασμό που να μπορούν όλοι να το δεχτούν. Αυτός είναι πάντα και ο ρόλος της εισηγήτριας. Αυτά τα γενικά τώρα, ε, επιμέρου. Θα πρέπει να το τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα ε, και σας είπα για ποιους λόγους για να το ε, ξεκινήσει αυτό η Σλοβακική Προεδρία στον τριμερή διάλογο. Βεβαίως θα τα ξανασυζητήσουμε από όλες τις πλευρές, από όλες τις σκοπιές, θα ακούσουμε και την Επιτροπή και το Συμβούλιο που εν μέρει μπορεί να διαφωνεί. Ε, ξέρουμε και τι λέει το Συμβούλιο και τι φρονεί σχετικά. Λοιπόν, εγώ αισιοδοξώ ότι θα καταλήξουμε σε μια καλή ε, εκδοχή που δεν θα περιορίζει καθόλου την κινητικότητα των εργαζομένων αλλά θα σέβεται κάποια πράγματα. Πολύ συγκεκριμένα λοιπόν σε αυτά που αναφέρατε για τον κύριο Μιζελία και τον Πέτερ Βαντάλεν. Δεν έχω να απαντήσω τίποτα. Η Κλάουδια Ταπαρντέλ και η Νέσα Γιάλα είπαν μερικά πράγματα που θέλουν απάντηση. Είπε η Κλάουδια ότι ορισμένες τροπολογίες είναι αντιφατικές. Ισχύει αυτό. Δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτές εξαιρέσει, αλλά γι' αυτό ήταν ε, για μένα δύσκολο με τις τροπολογίες των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Ορισμένοι ήθελαν οπωσδήποτε εξαιρέσει και άλλοι σε καμία περίπτωση. Προσπαθήσαμε να συγκεράσουμε και τις διάφορες κουλτούρες και τις παραδόσεις. Ας πούμε, Ρουμανία, Γαλλία, καμία σχέση. Ε, το καταλαβαίνω απολύτως και το σέβομαι. Αν θέλουμε όμως να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, ε, θα πρέπει να ταιριάζει όσο γίνεται σε όλους. Είπατε ότι χρειαζόμαστε ε, σαφείς κανόνες, μα υπάρχει το Συμβούλιο ΣΕΣΝΗ που είναι διεθνής οργανισμός και ε, έγκυρος, αλλά όχι αποκλειστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διεθνείς οργανισμούς και θεσμούς. Εκτός από τις ΕΣΝ υπάρχουν και άλλες επιτροπές, δεν είπαμε μόνο εκείνη. Και βεβαίως να υπάρχουν σαφείς κανόνες και προδιαγραφές. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 54 που με ρωτήσατε, είναι δική μου, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στο συμβιβασμό και υποθέτω ότι θα απορριφθεί Ορισμένοι ήθελαν και κάποιες τεχνικές προϋποθέσεις και έκαναν και τροπολογίες και δεν το θεωρούσα εγώ σωστό και το λέω και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τεχνικές απαιτήσει και πάντα είχα βάλει ανετικό πρόσημο ε, στον κατάλογο ψηφοφορία. Δεν εφαρμόζονται εδώ γιατί έχουν να κάνουν με κάποιε περιοχέ που στο παράρτημα αλλάζουν. Είναι πολύ τεχνικά αυτά τα θέματα και λεπτομέρειε και δεν το έκανα. Αυτά για την τροπολογία 54. Τι άλλο έχουμε. Α, Λοιπόν, την 54 τροπολογία λοιπόν Εκεί αναφέρθηκα σε χώρες που έχουν πλωτά ποτάμια και καταρτίζουν ναυτικούς ε, ε, και προτείνω μια εξαίρεση για χώρες όπως η Μάλτα που ακόμα δεν έχουν αρχίσει την εκπαίδευση αλλά μπορεί να την αρχίσουν. Για την 177 που ρώτησε η Νέσα για άλλα, 177 υπάρχει σε δύο συμβιβαστικές προτάσεις το πρώτο είναι στην συμβαστική 7 για το άρθρο 16 και το δεύτερο είναι στη συμβαστική 11. Έχω βάλει δύο νέες προτάσεις για το ότι έχει να κάνει με το ΣΕΣΝΗ για τις κατεξοδότηση και τις εφαρμοστικές πράξεις. Για λόγους έτσι, συνέπειας και συνοχής τα έχω βάλει εκεί και για το ε, πλαίσιο το νομικό για ε, ταχυγράφους ε, στα ποτάμια, ηλεκτρονικά το γράφουμε και αυτό. Ε, ο Βίμ είπε για την 20 ετία, τη μεταβατική περίοδο που είναι υπερβολική η χρονική περίοδος, βεβαίως δεν το έχουμε γράψει στους συμβιβασμούς για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκφράζει επιφυλάξεις. Τις φιλανδικές λίμνες τις έχουμε συμπεριλάβει. Και είναι μόνο για τη Φιλανδία και τίποτα άλλο. Κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους. Δεν βρίσκει εφαρμογή σε άλλες χώρες. Επίση είπαμε, κάτι που ισχύει τώρα, στι φιλανδικέ λίμνε υπάρχουν άνθρωποι που αρμενίζουν εκεί πέρα και έχουν εκπαίδευση μόνο για τι λίμνε αυτές και πουθενά αλλού. Και εφόσον δεν το κουνάνε από εκεί, καλά να κάνουν να έχουν αυτή τη φιλανδική κατάρτιση και να ταξιδεύουν μόνο στι λίμνε του. Αν έρχεται όμω ένα ναυτικό και λέει καλημέρα σα θέλω να πάω και στο Ρήνο, ε όχι, θα κάνει εκπαίδευση για το Ρήνο, γιατί δεν ξέρει να κυκλοφορεί στο Ρήνο. έχει ρεύματα, έχει ε, δυσκολίε τοπικέ. δεν μπορεί να έρθει από τη φιλανδική ε, λίμνη να κυκλοφορείς στο Ρήνο. Αυτά, ε, ως παράδειγμα, για να καταλάβουμε περί τίνο πρόκειται. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τη Φιλανδία, οφείλω να ομολογήσω. Σας είπα για τις τεχνικές απαιτήσει. Συμβαστική 14 υποθέτω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, αναφέρεται κυρίως στο τελευταίο σημείο που αφορά τη Γερμανία. Όταν είσαι ναυτόπες, δεν είσαι ναύτης, είσαι ακόμα κάτω από το ναύτη, ναυτόπες, ε, να έχεις μόνο επαγγελματική εμπειρία και να αρκεί αυτό να αναγνωρίζονται. Ε, ε, χωρίς ε, πτυχίο, χωρίς δίπλωμα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν περάσει θεωρητική εκπαίδευση, δεν μπορούν να δώσουν εξετάσεις. Το είπα στους συναδέλφους και το κατάλαβαν να παραμείνει έτσι. Και το υψηλό ποσοστό ατυχημάτων το έχω ακούσει κι εγώ από τον κλάδο, το έχουν υποστηρίξει πολλοί συνάδελφοι, γι' αυτό έχει παραμείνει στην πρότασή μας. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το διαχειριστεί κανεί. δεν ήθελα να φτιάξω εμπόδια ε, για να ε, υπάρχουν απαγορεύσεις στα ποτάμια, αλλά μπορεί ε, να είναι πρόβλημα κι αυτό. Αυτή είναι η θέση μας. Ψηφοφορία ελπίζω αύριο και όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στον τριμερή διάλογο. Θα έχουμε μεγάλη ευκαιρία και πολλέ δυνατότητες να το ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφοφορία αύριο λοιπόν, γιατί είχαμε γκρίνει την ημερήσια διάταξη. Ξέρω ότι υπάρχουν ε, διαφορές και ε, ο Πέτερ Φαντάλ το είπε έχουν υπέρ και κατά η αναβολή της ψηφοφορίας Έπρεπε τρει μέρε πριν να το είχατε ζητήσει, αν θέλετε αναβολή τη ψηφοφορία, αλλά παραμονή. Όχι, δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Θα ψηφίσουμε. Δεν μπορούμε να αναβάλουμε ούτε τη γενική ψηφοφορία, ούτε τη σειρά. Τελείωσε αυτό. Θα πρέπει να είμαστε συνεπεί. Αλλιώ ε, θα μπλέξουμε πολύ άσχημα και ζητώ συγγνώμη. Η ECR είναι μεγάλη πολιτική ομάδα και θα βρει κάποιον να στείλει να ψηφίσει. Δεν χάλασε ο κόσμος. Πάμε στο επόμενο θέμα. σε έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκον είναι έκθεση πρωτοβουλίας, συντάκτρια γνωμοδότησης δικιά μας είναι η κυρία Φώστερ, η οποία έχει και το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε και εσείς, είναι πρωτοβουλία από αυτή την Επιτροπή και έχουμε και γνωμοδοτήσεις από άλλες επιτροπές σχετικά για την πολιτική ανταγωνισμό και είναι μάλλον λυπηρό ε, το γεγονός πως τελευταία πρέπει να είμαστε πολύ μινιμαλιστές στις ε, γνωμοδοτήσεις μας και τελικά ούτε μισή σελίδα περιθώριο δεν μας δίνεται για τις απόψεις μας. Εν πάση περιπτώσει, ε, επειδή υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί, νομίζω πως χρειάστηκε να δείξουμε ιδιαίτερη αυτοπιθαρχία και να εστιάσουμε σε οκτώ ε, χώρους όπου έχουμε οκτώ συμβιβαστικές ε, τροπολογίες που καλύπτουν τα σημεία τα οποία είναι τα πιο σημαντικά σε σχέση με το θέμα του ανταγωνισμού. Η συνάντηση με τους κοιόδες ήταν πολύ επικοδομητική, έγινε στο Στρασβούργο και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για τον τρόπο με τον οποίο συνεισέφεραν στην όλη συζήτηση. Θα αναφερθώ εντάχει στα όσα συζητήσαμε με τους κιόδες και με τα όσα πιστεύουμε εμείς και θα ήθελα οι συνάδελφοι οι οποίοι ε, κάνουν πηγαδάκι μπροστά μου αν μπορούν να το διακόψουν. Sorry, it's just a bit off-putting. Okay, sorry. Συγχωρείτε γιατί πραγματικά ε, χάνω την, ε, το συνειρμό μου. Λοιπόν, συμβιβαστικές τροπολογίες εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και διασυνδεσιμότητα. Ε, δεύτερον, η κακή εφαρμογή και επιβολή της πολιτικής για τις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαντικό και αυτό. Μία τροπολογία για την απομάκρυνση των κανονιστικών, ρυθμιστικών και πραγματικών εμποδίων. Μετά μιλήσαμε για την ψηφιακή πολιτική και για την ε, οικονομία του διαμοιρασμού και μετά μιλήσαμε για τις εξωτερικές συμφωνίες αεροπλοείας, κάτι το οποίο συζητήσαμε αρκετά σήμερα το πρωί στα πλαίσια της στρατηγικής για την αεροπλοεία, οπότε καταλαβαίνετε πως είναι ένα θέμα το οποίο διέπει αρκετές τροπολογίες. Κατόπιν μιλήσαμε για θέματα ανταγωνισμού ε, και κάποιες ε, καταστάσεις οι οποίες προέκυψαν που ήταν μάλλον απογοητευτικές και για το τέταρτο πακέτο για τους σιδηροδρόμους ξέρουμε πως αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί εκεί μια τροπολογία λοιπόν συμβαστική και τέλος μια αντίστοιχα για τον τουρισμό για την πρώτη συμβαστική τροπολογία εμβάθυνση της ε, ενιαίας αγοράς και διασύνδεση μότητα βεβαίως θα πρέπει να έχουμε ίσους κανόνες παιχνιδιού για όλους, αλλά να σεβαστούμε και τις αρχές της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ συμπεριλαμβάνουμε και την κοινωνική διάσταση. Έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πως η αγορά αυτή θα λειτουργεί ομαλά. Τονίσαμε πάρα πολύ τη σημασία διασυνδεσιμότητας και των δομών ε, συγκοινωνιών και μεταφοράς, όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη και την προσφορά υπηρεσιών δημοσίων και ιδιωτικών σε περιφέρειες και σε κέντρα. Άρα λοιπόν και εδώ την περιφερειακή πολιτική τώρα για την ε, αδύναμη επιβολή, να σας πω πως υπάρχει σφαιρική και πλήρης νομοθεσία, την οποία έχουμε αποκτήσει σιγά σιγά με τα χρόνια και παρόλα αυτά υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δεν εφαρμόζουν νομοθεσία της δικής μας Επιτροπής, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί. Είναι σαφής και δεν μιλώ για κατάσταση όπου ξέρουμε πως έχουμε κάποια κάποιες καθυστερήσεις για περίπλοκους λόγους, αλλά για ε, παράδειγμα νομοθεσία η οποία ισχύει ήδη στα κράτη-μέλη και δυστυχώς είναι αρκετά συχνό η νομοθεσία αυτή να μην εφαρμόζεται. Και αυτό δεν το αντιμετωπίζουμε με κάποιο τρόπο. Επίσης αναφέρθηκα στις καταναλωτές και για να εξασφαλίσουμε πως όλα λειτουργούν σωστά, να σας πω πως χρειάζεται αυτό έτσι ώστε η αγορά να λειτουργεί για όλους και για τους εργαζομένους και για τους καταναλωτές και για το περιβάλλον και για τη βιομηχανία, και για την, τον επιχειρηματικό κόσμο. Άρα λοιπόν κάνουμε μία αναφορά εδώ στους εργαζομένους και στο περιβάλλον. Ε, φυσικά, τεχνητά και κανονιστικά εμπόδια. Και εδώ πάλι όταν μιλάμε για φυσικά εμπόδια υπάρχουν λόγια για τους οποίους δεν μπορούμε να μετακινηθούμε από μέρος σε μέρος. Φυσικά εμπόδια. Τώρα, έχουμε πολλές φορές και ακατάλληλη νομοθεσία όπου μπορεί να υπάρχει, για παράδειγμα, ε, επιτόπου τοπική νομοθεσία που δεν μας επιτρέπει να ακολουθήσουμε μια κοινή προσέγγιση και αυτό θα πρέπει να το δουν τα κράτη-μέλη. Θέλουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε πως θα διευκολύνουμε την κινητικότητα, τη διασυνοριακή, όπως επίσης και την εδαφική συνεργασία. Για το λόγο αυτό προφανώς υπογράψαμε όλη την ενιαία αγορά. Και όλα αυτά θα ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό. Παρακάτω λοιπόν, συνεργασία, ψηφιακές τεχνολογίες. Τόσα χρόνια καθόμαστε εδώ και συζητάμε για τις ευφυείς συγκοινωνίες, ε, ναυσιπλοεία, αεροπλοεία, γαλιλαίο, ε, GNSS, όλες αυτές οι έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακές τεχνολογίες οι οποίες πραγματικά έχουν κατακλείσει τον κόσμο και ήμασταν πολύ επικοδομητικοί πολλές φορές όταν έχουμε εργαστεί εμείς παράλληλα με την Επιτροπή Ήτρε. Άρα λοιπόν εδώ απλώς τονίζουμε ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τη συνεργασία αυτή γιατί προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα στους κλάδους και παρόλα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως το νομικό πλαίσιο είναι αρκετά ξεκάθαρο έτσι ώστε να χρησιμοποιούμε τα πλονεκτήματα που προσφέρει χωρίς υπερβολική ε, νομοθετική προσπάθεια. Τώρα για τις εξωτερικές ε, συμφωνίες για την αεροπλοεία δεν θα πω κάτι παραπάνω από ό,τι ακούσαμε το πρωί, τα είπε και ο Πάβελ. Και πρέπει να σου πω ότι ιστορικά αυτός ο κλάδος αποτελεί έναν με πάρα πολύ ε, σκληρή και αυστηρή νομοθεσία. Το χρειάζεται. Οι θέσει εργασία είναι υψηλή ποιότητας, τα πρότυπα ασφαλεία είναι πάρα πολύ αυστηρά και λαμβάνουμε υπόψη και τα δικαιώματα των εργαζομένων στον κλάδο, γιατί θα πρέπει να είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι και τονίζουμε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λόγο όταν μιλάμε για αυτέ τι εξωτερικέ συμφωνίε, έτσι ώστε να είναι κατάλληλες και βέβαια θυμητός ανταγωνισμός, ίσοι κανόνες για όλους. Τα αναφέρουμε και πάλι. Τώρα για τις οδικές μεταφορές, εδώ το κλειδί για το συμβιβασμό ήταν να βρούμε κάποιο τρόπο, στηρίζοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να δούμε τα μέτρα τα οποία λάβαμε κάποτε και καταδικάζουμε το γεγονός πως κάποια κράτη-μέλη πως κάπνουν την ενιαία αγορά. Δεν χρειάζεται να πω σε λεπτομέρειες, τα γνωρίζουμε όλοι αλλά δεν λειτουργεί έτσι η αγορά και ούτε ήταν αυτό ο στόχο της. Δηλαδή δεν μπορεί μια ιδέα ενό κράτου μέλου να διακυβεύει τις οδικέ διασυνοριακές μεταφορές. Τέταρτο πακέτο σιδηροδρόμων. Θέλουμε να κλείσει αυτό το θέμα το συντομότερο και βέβαια η έγκριση και του τεχνικού πυλώνα που χρειαζόμαστε όλοι. Επίσης έχουμε ειδικά ε, κυρία Νταμποντέλ, την τροπολογία 8. Ελπίζω για τον τουρισμό αυτό που συντάξαμε να είναι ικανοποιητικό, γιατί εστιάζει περισσότερο στις συγκοινωνίες και βέβαια ξέρετε πως ο τουρισμός για την αλυσίδα διανομής είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Σε γενικές γραμμές λοιπόν αυτή την προσέγγιση ακολουθούμε, είναι σύντομο, είναι συνεκτικό, είναι δυσέλιδο και ελπίζω πως η Επιτροπή θα το δεχθεί ως έχει. Εστιάζει πάρα πολύ στις συγκοινωνίες. Ευχαριστώ τους Κιώδης και όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την κυρία Φώστερ γιατί πρέπει να σας πω πως αυτές οι οκτώ τροπολογίες αποτελούν απόρρια πολύ ισορροπημένης προσπάθειας και εργασίας. Τα κεντρικά ζητήματα τα οποία θέσατε βρίσκονται εδώ στον κατάλογο που μας δώσατε αριθμημένα και θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις για κάποιες λεπτομέρειες με τις οποίες εμείς ε, δεν μπορούμε να ε, συμφωνήσουμε πάντα. Αέρο, μεταφορές, σιδηροδρομικές μεταφορές, τέταρτο πακέτο, δικές μεταφορές, αεροπλοεία. Όλα αυτά τα θίξαμε σε γενικές γραμμές και μιλήσαμε για τις διάφορες πτυχές της ενιαίας αγοράς. Έχουμε όμως τα λιμάνια. Τα λιμάνια δεν τα συμπεριλάβαμε στις τροπολογίες. Ξέρετε πως τον κανονισμό για τα λιμάνια θα τον ψηφίσουμε σύντομα και λυπάμαι που δεν υπάρχει τροπολογία που να ασχολείται με την ε, πολιτική μας για τα λιμάνια. Βέβαια δεν είναι κάτι που ενοχλεί ιδιαίτερα γιατί το καινούριο κανονισμό δεν μπορώ να σας πω πως τον στηρίζω ένθερμα ούτε πως με ενθουσιάζει. Είναι βέβαια προϊόν της εργασίας των συναδέλφων, αλλά δεν σας κρύβω πως έχουμε και μια τροπολογία την οποία θα υποβάλω ε, σύντομα, γιατί στον κανονισμό για τα λιμάνια υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν με ικανοποιούν. Για παράδειγμα, ανταγωνισμός και διαφάνεια δεν θίγονται επαρκώς, λιμενικές υπηρεσίες. Τα έχω πει και προσπάθησα να το τονίσω αυτό όταν ψηφίσαμε τον κανονισμό. Ε, πάντως προσπαθώ να τα ξαναδούμε μέσω των τροπολογιών. Επίσης, κρατικές ενισχύσεις και εκεί έχω προτείνει μια τροπολογία και θα ήθελα να υπενθυμίσω πως έχουμε υπερβολικά πολλές διαφορές μεταξύ όσων θεωρούν κρατικές ενισχύσεις στις μεταφορές στα κράτη-μέλη. Η κυρία Φώστερ μας το υπενθύμισε. Έχουμε την ενιαία αγορά. Θα πρέπει να ισχύει με τον ίδιο τρόπο για όλους. Και τέλος, για τα σημεία αυτά, να σας πω ότι έχουμε ακόμα δύο τροπολογίες ε, και κάποιες σκέψεις για τα ε, χρηματοδοτικά εργαλεία. Για παράδειγμα, ε, το ΣΥΦ και το ΕΦΣΥ. Θα ακούσουμε βέβαια αργότερα τον Επίτροπο κύριο Κατάινεν για να μας πει τι θα γίνει με το πακέτο, πακέτο Juncker 2.0 και νομίζω πως σύντομα ε, θα ληφθούν υπόψη αυτά τα οποία προτείνουμε. Για να καταλήξω στο συμπέρασμά μου, συγχαρητήρια στη συνάδελφα, ήταν πολύ ισορροπημένη προσπάθεια που έκανε. Αλλά βέβαια, ω σύνοψη πρέπει να σας πω πως είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε με κάτι το οποίο είναι τόσο ολιγόλογο πάντα. Για τις επενδύσεις. Για τις επενδύσεις. Νομίζω θα έπρεπε να έχουμε συμπληρώσει περισσότερα. Έχουμε πει πολλά για το περιβάλλον, για την κοινωνική διάσταση. Δεν θα πρέπει όμως να χάνουμε καμία ευκαιρία που μας δίνεται έτσι ώστε να έχουμε μια ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων, των αμέτρητων απαιτήσεων που έχουμε για να έχουμε μια σωστή πολιτική επενδύσεων και παράλληλα για να εξυπηρετήσουμε τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς μας στόχους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κλάουντια Ταπάρντελ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για την Επιτροπή Μεταφορών η παρούσα γνωμοδότηση. Εδώ έχουμε την ευκαιρία να εξηγήσουμε στους συναδέλφους της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων ποιες είναι οι δικές μας προτεραιότητες για τις μεταφορές στην Ευρώπη και ιδιαίτερα για τον ανταγωνισμό. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ εδώ την κυρία Φώστερ για τη δουλειά της και επίση για την προθυμία της. Ήταν πάντα διαθέσιμη να μας ακούει και τις δικές μας θέσεις των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Τι λέμε λοιπόν εμείς, ότι θέλουμε να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα του κλάδου και της βιομηχανίας αλλά και τις κοινωνικές ε, ε, πτυχές. Γενικά τα έχουμε καταφέρει, υπάρχουν κάποιες σημαντικές ε, τροπολογίες για πολύ κρίσιμα θέματα όπως είναι η κοινωνική προστασία, η είσοδος νέων φορέων στη νέα μορφή συμμετοχική οικονομίας και τις οδικές μεταφορές επίσης. Οι συμβαστικές τροπολογίες μας βρίσκουν σύμφωνους σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να καταλήξουμε για τα σημεία 5 και 6 οριστικά σήμερα. Υπάρχουν δυνατότητες. Ε, τα κοινωνικά ζητήματα θα θέλαμε να τονίζονται λίγο περισσότερο, ε, δηλαδή τροπολογίες 1 και 9 της κυρίας Γεβόνταλόν θα πρέπει να ψηφιστούν χωριστά. Όπως επίσης και η τροπολογία παριθμών 16 που αναφέρεται στη συμβαστική 6. Παρακαλούμε χωριστή ψηφοφορία. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ. Ήταν εξαιρετική συνεργασία μας. Και είναι πάρα πολύ καλή γνωμοδότηση. Ευχαριστώ ο κύριος Τελίτσκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συνταχθώ και εγώ με τους συναδέλφους και να συγχαρώ την εισηγητρία για τη δουλειά που έκανε και στην ε, διατύπωση και στην σύνταξη και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε στη συναντήση με τους σκιώδες. Πρέπει να πω πως το σχέδιο κειμένου μου αρέσει και μου αρέσουν και τα αποτελέσματα. Αρκετές τροπολογίες ελήφθησαν υπόψη. Νομίζω λοιπόν πως βρήκαμε μια σωστή ισορροπία και αυτό το πετύχαμε από την αρχή. Όπως και στα πλαίσια της στρατηγικής, έτσι και εδώ θεωρώ πως παρόλο που είναι σύντομο το κείμενο, έτσι πρέπει να είναι, είναι κατάλληλο το κείμενο γιατί δίνει το σωστό μήνυμα και πρέπει να πω ότι το συμπεριλαμβάνει όλα. Στο πυρήνα βρίσκεται η εσωτερική αγορά και βεβαίως το μήνυμα είναι ότι δεν μπορούν κάποια κράτη-μέλη μέσω κάποιων δραστηριοτήτων να παρακολύουν την ενιαία αγορά και νομίζω ότι η διατύπωση που διαλέξαμε είναι καλύτερη και μια καλή ισορροπία μεταξύ μιας απλουστευμένης ε, δυνατότητας ε, επενδύσεων που παράλληλα προστατεύει τα κοινωνικά πρότυπα που έχουμε. Πριν μπω λοιπόν σε υπερβολικές λεπτομέρειες, να σας πω πως ε, μας εξηγήθηκαν οι τροπολογίες, οι συμβαστικές τροπολογίες και εγώ θα συστήσω στην, στους φιλελεύθερους να υπερψηφίσουν. Ξέρω ότι έχουμε κανένα δύο σημεία τριβής. Και ίσως κάποιοι θεωρούν πως οι τροπολογίες τους δεν ελήφθησαν δεόντως υπόψη, αλλά ξέρουμε όμως ποιος είναι ο κίνδυνος εκεί. Και επειδή είναι ισορροπημένο εδώ το κείμενο, θα πρέπει να προσπαθήσουμε κι εμείς έτσι ώστε να μην αλλάξουμε το νόημα του κειμένου μέσω υπερβολικό, υπερβολικό αριθμού τροπολογιών. Εν πάση περιπτώσει, ας παραμείνουμε εκεί στο ελάχιστο για τις ξεχωριστές πληροφορι... ε, ψηφοφορίες, με συγχωρείτε, και να στηρίξουμε ένα σχέδιο κειμένου που είναι πολύ καλό και που στέλνει το σωστό μήνυμα. Όχι μόνο στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, αλλά στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ η Μαρία Κίλωνεν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω, συνάδελφε, για το κείμενο αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο ε, στο Κοινοβούλιο πολλές φορές έχει φέρει ρήξεις, πολλές φορές είναι τελείως διαφορετικές οι απόψεις μας, αλλά η δική σας προσέγγιση ήταν πολύ επικοδομητική. Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με όλες τις συμβιβαστικές προτάσεις, αλλά αυτό είναι κομμάτι της πολιτικής ζωής είναι διεθνής η φύση της, ε, των μεταφορών, είναι τα logistics, είναι ο τουρισμός, είναι ο ανταγωνισμός που είναι και διασυνοριακός, η αεροπλοεία, ε, ο ανταγωνισμός μεταξύ Ευρώπης και τρίτων χωρών και ίσως αυτή η προστατευτική προσέγγιση για να προστατευτούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες εδώ στην Ευρώπη να είναι προβληματική. Τώρα η αυτή η πατάτα στις οδικές μεταφορές είναι η προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων και το πώς συνδυάζουμε τα όσα κάνουμε σε χώρες που αυτά κοστίζουν λιγότερο, όπως οι άλλες κοστίζουν περισσότερο. Τώρα για το σιδηροδρομικό πακέτο, να σας πω πως η αγορά εκεί χτίστηκε με εταιρείε οι οποίες είχαν μια, ένα φυσικό μονοπόλιο το οποίο αυτή τη στιγμή εμείς ε, αποξηλώνουμε και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δημιουργεί αναταραχές. Οι διάφορες ε, δυνατότητες μεταφορών ανταγωνίζονται για ποιον καταναλωτή θα αρπάξουν. Ε, έχουμε την ψηφιοποίηση η οποία έχει φέρει την επανάσταση στον χώρο των μεταφορών. Έχουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ εταιριών εταιριών οι οποίες είναι χρόνια στον κλάδο και των νεοεισερχομένων και βέβαια θα πρέπει να δούμε και υπό ποιες προϋποθέσεις στον κλάδο αυτό θα επιβιώσουν κάποιοι. Δεν νομίζω πως θα μπορούμε να βλέπουμε τον ανταγωνισμό ως ένα, μια γρήγορη λύση που θα οδηγήσει είτε στην ευτυχία είτε θα μας καταδικάσει στην καταστροφή. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως το νομοθετικό πλαίσιο για όλες τις συγκοινωνίες και μεταφορές θα είναι ξεκάθαρο και όλες οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίζονται με ισότιμο τρόπο. Πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε πως όλος ο κλάδος των μεταφορών υπάρχει υπάρχει για να υπάρχει κινητικότητα και μπορούμε να μεταφέρουμε πολίτες, ε, επιβάτες, εταιρίες, αγαθά ε, σε διάφορους τόπους. Στην απόφαση που θα πάρουμε ας θυμόμαστε πως όλοι οι κανόνες έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τον τελικό καταναλωτή έτσι ώστε να του προσφέρουμε την καλύτερη δυνατόν εναλλακτική. Πήγαμε και επισκεφθήκαμε την Ιαπωνία και εκεί μου υπενθύμησαν πως η προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη ε, πιο πολύ από όλα τα συμφέροντα του καταναλωτή είναι αυτή η οποία τελικά κάνει τη διαφορά. Και εκεί είναι πολύ η υγιής η αντιμετώπιση τους για ολόκληρο τον κλάδο, όπου θέλουν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες όσο το δυνατόν καλύτερα και ξέρετε πως οι Ευρωπαίοι πολλά θα είχαμε να διδαχτούμε. Ευχαριστώ πολύ η Marie-Christine Αρνοτζού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Φώστερ. Είναι πάντα ενδιαφέρον και πολύ επικοδομητικό το έργο της, ακόμα και αν διαφωνούμε βαθιά για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ως ε, Γαλλίδα βουλευτής, εγώ διαπιστώνω ότι ελεύθερος ανταγωνισμός και ο πρόσκοπτος που ε, υπόσχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μία χήμερα και κάθε μέρα χάνονται θέσεις εργασίας, καταργούνται, ισοπεδώνονται οι κοινωνικές προστασίες και ασφάλεια. Ο κλάδος των μεταφορών ε, είναι παράδειγμα χαρακτηριστικό και θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό στη γνωμοδότησή μας προς την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Στη Γαλλία οι πολιτικές των Βρυξελών ήταν ολιγοπολαίθριες. Ο ευρωπαϊκός ανταγωνισμός οδήγησε στο να χαθούν σχεδόν τελείως οι Γάλλοι ε, οδηγοί φορτηγών που έχουν αντικατασταθεί από φτηνούς ξένους ε, που τρίβουν τα χέρια τους οι εταιρείε που δεν έχουν και ε, μεγάλο ενδιαφέρον για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Είναι αντίστοιχο αυτό φαινόμενο των σημαίων ευκαιρίας. Υπάρχει λοιπόν και στις θαλάσσιες μεταφορές και στις αερομεταφορές με το χαμηλό τόξο, κόστος υπό την πρόφαση ότι είναι υπέρ των ε, επιβατών που θεωρούνται μόνο καταναλωτές. Τι να σκεφτεί κανείς για τις ξένες συμμετοχές σε πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες, η Αλιτάλια που την αγόρασε το κατά, η ε, τα XPO ε, ε, κάνουν αντίστοιχα, το λιμάνι του Πειραιά το γόρασε η Κινέζικη Κόσκο κτλ. Άρα καταστρέφουμε στρατηγικές υποδομές, θέσεις εργασίας, παραχωρούμε στρατηγικές υποδομές ε, ξεπουλάμε ε, τις ευρωπαϊκές αξίες. Το όνομα ε, της ανταγωνιστικότητας και της αποδυτικότητας έχουμε αφήσει στη μοίρα της και τη χωροταξία. Στη Γαλλία δεν γίνεται πουθενά πια καθόλου χωροτακτικό σχεδιασμός. Και ειλικρινά μια τέτοια πολιτική ανταγωνισμού είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν συμπεριλάβατε καμία από τις δικές μας τροπολογίες στο συμβιβασμό. Παράδειγμα, να σας αναφέρω μία μερικές δηλαδή, όχι μόνο μία, όπου ζητούσαμε ενδεχόμενες εξωτερικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνονται ε, με ε, πλήρη διαφάνεια τουλάχιστον από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Ισαπέλα Τεμόντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρεμβαίνω για να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους και για τη δουλειά τους που ήταν άριστη, όπως είπε και η συγκήτρια, ακόμη και ως προς τους χαρακτήρες που προβλέπονται για να καλύψει ένα θέμα τόσο ευρύ όπως ανταγωνιστικότητα κανείς δεν είναι αρκετή. Όμως νομίζω ότι χάρη και στις τροπολογίες που είναι σκοπιμότατες και στοχές θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στο σωσή ισορροπία. Θέλω να αναφερθώ στη συνεργατική οικονομία. Το στοιχείο αυτό που προβλέφθηκε και είναι σημαντικό γιατί το βλέπει και η Επιτροπή Εξωτερικής Αγοράς και εκεί θα υπάρξουν και οι σχετικές νομοδοτήσεις από εμάς, οπότε καλό είναι να αρχίσουμε από τώρα να βλέπουμε το θέμα και να εκφράζουμε τις απόψεις μας. Και για άλλα σημεία θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που δέχτηκε κάποιες από τις παρατηρήσεις μας, όλο ιδιαίτερα στη βελτίωση των, συνθηκών, των κοινωνικών συνθηκών για τους εργαζομένους και τα πρότυπα ασφάλειας καθώς και την βελτίωση για τον σιδηροδρομικό κλάδο και την ε, ε, απάλληψη των τεχνικών φραγμών με την δέσμη μέτρων για τους ιδεοδρόμους. Πραγματικά αυτό ήταν πολύ σκόπιμο, διότι υπάρχει μόνο ένα μέρος για τον τουρισμό, αναγνωρίζοντα ότι είναι μια σημαντική συνιστόσα της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόληση. Γι' αυτό λοιπόν και πάλι ευχαριστίε προ όλου για αυτή την πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Μάρεξ Σταβινό από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Good morning, Phil Roberts. Καλημέρα σας, είμαι από την ε, DG Move και δεν είμαι ο Μάρεκ, ο Μάρεκ κάθεται δίπλα μου. Θα ήθελα να μιλήσω και για την έκθεση και τις τροπολογίες. Δεν έχουμε δει τις συμβιβαστικές τροπολογίες ακόμα, οπότε είναι πολύ δύσκολο να τις σχολιάσω πιο συγκεκριμένα, αλλά ακούσαμε πολύ προσεκτικά τα όσα σχολιάσατε σήμερα το πρωί και πολλές από τις τροπολογίες μπορούμε να τις δεχτούμε, γιατί είναι πολύ ισορροπημένη αυτή η γνωμοδότηση. Η κυρία Φώστερ, όπως πάντα στην έκθεσή της, ήταν πολύ συγκεκριμένη, ασχολήθηκε αυστηρά με το θέμα που είχε μπροστά τη και όπω είπαμε τη συζήτηση τον περασμένο μήνα, είναι καλή έκθεση γενικά. Την καλωσορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν τόσα πολλά τα θέματα που έθεσε για τι μεταφορέ, που ήταν πολύ δύσκολο για κάθε τροπολογία να σχολιάσουμε. Όμω είναι κάποια σημεία κυρίω για το πακέτο για τι οδικέ μεταφορέ που μιλήσαμε για τον ανταγωνισμό Έχω τον κύριο Ράσμουσεν που είναι ο εμπειρογνώμονά μου και ο οποίο θα μπορέσει να σχολιάσει κάποια από τα θέματα τα οποία θίξατε. Ευχαριστώ. Όπως είπε και ο Φιλ, Καταρχήν είναι πολύ θετικό πως κατάφερε να καταλήξει σε συμβαστικές τροπολογίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί δείτε τι γίνεται με τα κράτη-μέλη. Εκεί υπάρχει εξαιρετική πόλωση των απόψεων και φαίνεται να είναι αρκετά δύσκολο να καταλήξουμε σε ένα είδος ε, συμβιβασμού. Τουλάχιστον όπως έχουν τα πράγματα σήμερα. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προετοιμάζει αυτές τις πρωτοβουλίες για τις οδικές μεταφορές, όπου θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία, όπως έκανε και η Επιτροπή Μεταφορών. Βέβαια υπάρχουν τα μέτρα για την ενιαία αγορά, έχουμε την πρόσβαση στην αγορά, την πρόσβαση στο επάγγελμα και εδώ συμπεριλαμβάνουμε και το καμποτάζ, αλλά υπάρχει και η κοινωνική διάσταση και τα ζητήματα αυτά τα οποία συζητιούνται πολύ σήμερα και θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να φέρουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των δύο ομάδων κρατών, ε, γιατί, επαναλαμβάνω, επικρατεί αρκετή πόλωση. Πιο πολλές λεπτομέρειες για αυτά που εξετάζουμε. Για το καμποντάζ, για παράδειγμα, είναι ένα εξαιρετικά κανθόδε ζήτημα, Εκεί δεν έχετε εσείς συμβασική τροπολογία, αλλά είναι ήδη τροπολογία, οπότε γι' αυτό το θίγω. Εκεί πιστεύουμε πως χρειάζεται να ε, κινηθούμε προσεκτικά και να είμαστε και πολύ σαφείς για το ποιοι είναι οι κανόνες. Έτσι ώστε να επιβάλλονται οι κανόνες, γιατί νομίζω ότι η επιβολή των κανόνων είναι ένα από τα σημεία ε, στα οποία στάθηκε πολύ συχνά η Επιτροπή Μεταφορών. Τώρα, αν δεν υπάρχουν πιο συγκεκριμένα ερωτήματα, δεν θα μπω εδώ σε πιο πολλές λεπτομέρειες. Πάντως, επειδή βρέθηκε ο συμβιβασμός και η ισορροπία, πιστεύω πως πήγαμε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, καλό θα είναι να μου δίνετε τις σωστές πληροφορίες προηγουμένως για να μην δίνω το λόγο σε λάθος άνθρωπο. Για το μέλλον αυτά, για να τα ρυθμίσουμε τη θαυμάσια και τώρα ξανά το λόγο η Τζάκη Φώστερ. much. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τους σκιώδει ηγητέ για τι τόσο επικοδομητικές τους παρατηρήσεις. Θα ήθελα να πω πω πολύ συχνά, και αυτό ισχύει για όλους από εμά, όταν περιοριζόμαστε στο χώρο που έχουμε διαθέσιμο και χρειάζεται να συμβιβαστούμε, δεν φτάνουμε πάντοτε στο κατάλληλο μείγμα, γιατί πολλές φορές χωρί να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε απαραίτητα, οι τροπολογίε δεν είναι οι κατάλληλε. Και γι' αυτό θα γίνουν και αρκετέ ξεχωριστέ ψηφοφορίε και νομίζω ότι εκεί οι συνάδελφοι θα καταφέρουν να στηρίξουν ή να μην στηρίξουν αυτά τα οποία ε, συζητάμε. Πάντως, όποιος και να είναι εισηγητής, οι τροπολογίες που συχνά ε, υποβάλλουμε προσθέτουν Και το κείμενο που έχουμε είναι πολύ συμπυκνωμένο. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, ακριβώς επειδή δεν είχαμε χώρο και χρόνο, είναι πολύ ε, επικεντρωμένο σε αυτά που μας αφορούν. Ξέρω ότι κάποιες ομάδες ε, είχαν κάποια ζητήματα, ένα, δύο τα, θα τα ψηφίσουμε ξεχωριστά, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις οι τροπολογίες που ζήτησαν να μπουν στο συμβιβασμό δεν τέριαζαν. Θα είχαν αλλάξει ολόκληρο το πακέτο αυτό το συμβιβαστικό. Τώρα, κύριε Σαλίνη, πολύ σωστά μιλήσατε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και για τους περιορισμούς που αντιμετωπίσαμε. Εμείς δεν μπορούμε κάθε φορά να συμπεριλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια και προσπάθησα να επικεντρώσω σε μια διαφορετική, ελάχιστα διαφορετική οπτική γωνία κάποια στιγμή τώρα για τις επενδύσεις. Εάν δεν έχουμε επενδύσεις δεν θα έχουμε πλέον κλάδο μεταφορών. Οπότε, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Πάντα προσπαθούμε να ε, προσελκύσουμε καλέ στήρες επενδύσεις, ναι. Τώρα για τα λιμάνια, κοιτάξτε, τρεις φορές το έχω ζήσει το έργο. Και ακόμα πρέπει να σας πω πως είμαι ζωντανή. Γιατί το 2000 ξεκινήσαμε τον κύριο Φλέκενστάιν τον καημένο. Και πρέπει να σας πω, αν αυτό σα κάνει αισθάνεστε καλύτερα, εγώ για τα λιμάνια δεν στήριξα τον κανονισμό. Όμω η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου τον στήριξε και τώρα πρέπει το θέμα αυτό επιτέλου να κλείσει γιατί απελευθερώσαμε τα λιμάνια στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από 35 χρόνια τα ιδιωτικοποιήσαμε. Οπότε γι' αυτό δεν το ανέφερα, γιατί νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει μέχρι θανάτου το θέμα. Μεγάλος φάκελος που ελπίζω πως έχει κλείσει πια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Κλάουδια. Ναι, ήταν σημαντικό να μιλήσουμε για τον τουρισμό, γιατί έχει να κάνει με την αλυσίδα ανεφοδιασμού και πολλής ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου μεταφορών εξαρτάται από τον τουρισμό. Θέλουμε, θέλουμε να στηρίξουμε αυτούς που ταξιδεύουν είτε για επιχειρηματική δραστηριότητα είτε για αναψυχή. Πάβελ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και του υπόλοιπου συναδέλφου. Πετύχαμε μια καλή ισορροπία και συμφωνώ. Συμφωνώ με την παρατήρηση πως πολύ συχνά συμφωνούμε να διαφωνήσουμε, αλλά το κάνουμε πάντα με ευχάριστο τρόπο. Και γι' αυτό πρέπει να σπανίκουμε και σε διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Πάντως ναι, δέχτηκα αρκετές από τις παρατηρήσεις, τις έλαβα υπόψη. Και στη Μαρή Κριστίν, την καλή μου φίλη, ήθελα να πω το εξή. Μιλήσατε για τους οδηγούς, τους Γάλλους οδηγούς. Και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε αντιπαράθεση εδώ για το αν είναι Βρετανοί ή Γάλλοι οδηγοί, αλλά σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ, όταν ήμουν 21, πήγα να δουλέψω σε μια εταιρεία που ήταν η British Airways και ήταν στην νηπιακή κατάσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η καλύτερη μου φίλη από τότε είναι η Ολλανδή, η οποία είχε έρθει από την Ολλανδία και ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να δουλέψει σε αυτή την καταπληκτική εταιρεία. Και πολλοί συνάδελφοι από τότε ήταν Γάλλοι. Και είχαμε και μέλη πληρώματος που ήταν από την Πολωνία, από τη Γερμανία και η εταιρεία για την οποία τότε δούλευα είμαι περήφανη να πω πως ήταν πραγματικά προοδευτική γιατί ως ε, ως αεροπορική εταιρεία έλεγε πως δεν ζεις μέσα σε ένα κενό για να είναι επιτυχημένη η εταιρεία σου στον κλάδο των μεταφορών θα πρέπει να καλωσορίζεις όλους τους νέους ερχόμενους γιατί προσφέρουν προστιθέμενη αξία. Και νομίζω ότι ήταν μια εταιρεία που πραγματικά ήταν πολύ επιτυχημένη. Άρα λοιπόν λαμβάνω υπόψη τα όσα είπες για τους οδηγούς οι οποίοι δεν πληρώνονται όπως όσο θα έπρεπε ή όπου οι αλλοδαποί, οι οδηγοί ίσως πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Είναι δίκαια αυτή η παρατήρηση και γι' αυτό το λόγο ήθελα να θίξω το θέμα της επιβολής και η επιβολή της εργασιακής νομοθεσίας είναι αρμοδιότητα του κράτους μέλους. Οπότε Εάν υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πέφτουν θύματα εκμετάλλευση σε κράτη-μέλη, υπάρχει εκεί εργασία και νομοθεσία και ευρωπαϊκή και εθνική. Άρα λοιπόν είναι δική τους ευθύνη να εξασφαλίσουν πως ε, πραγματικά θα πατάξουν το φαινόμενο αυτό των επιχειρήσεων που πολλές φορές εκμεταλλεύονται εργαζομένους. Γιατί σίγουρα εγώ δεν μπορώ να δεχτώ κάτι τέτοιο, γιατί εγώ προέρχομαι από τα συνδικάτα, ξέρετε. 15 χρόνια ήμουνα ε, συνδικαλίστρια. Οπότε το είπα για να σου απαντήσω, αλλά πέραν αυτού είμαστε διεθνείς. Είμαστε η καταπληκτική Ευρωπαϊκή Ήπειρος και πάντα μέσα στην Ευρώπη είχαμε μετακινήσεις και νομίζω ότι όλους μας έχει ωφελήσει αυτό. Για το λόγο λοιπόν τούτο, εγώ έχω αυτές τις τροπολογίες και δεν είναι προσωπικό και γι' αυτό όποτε θες μπορούμε να πιούμε ένα καφέ και να τα συζητήσουμε γιατί έτσι πρέπει να είναι η πολιτική. And uh, we're very happy for it to go. Ευχαριστώ πολύ και θα χαρώ πολύ που θα περάσει το θέμα αυτό από την ψηφοφορία. Αν μας υπερψηφίσουν, που δεν προδικάζω, είναι μια καλή γνωμοδότηση για να την αναλάβει και η ΕΚΟΝ, γιατί νομίζω ότι αποτελεί αναπόσταστο τμήμα της δικής τους έκθεσης και δεν νομίζω ότι έχουν καμία δικαιολογία να μας πούν ότι η δική μας γνωμοδότηση δεν ταιριάζει στη βασική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Και η δική μου εμπειρία είναι ότι ωραίοι άνθρωποι κάνουν και ωραία σχόλια. Äh, Αύριο είναι η ψηφοφορία. Τώρα θα πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα. Διότι η ειδική ομάδα για το τουρισμό θα έρθει στις 11 ε, και 4. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι ενδεικτική η χρόνη στην ημερήσια διάταξη. Εκτιμήσει κάνουμε. Μην το δένετε κιόλα, Δηλαδή ότι ε, θα πρέπει να έρθουν 11 και 4. Ορίστε, καμιά φορά τελειώνουμε και νωρίτερα. Παρακαλώ το λαμβάνουμε υπόψη. Υποχρεωτικό διάλειμμα λίγων λεπτών. Και πολλών μάλιστα, γιατί έχουμε δύο προσκεκλημένους. 11 και 4 συνεχίζεται. Η δική ομάδα για το τουρισμό. Mr. President, we have a translation problem with Romanian, so we don't hear in our headsets Romanian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 Ε, νομίζω ότι μπορούμε τώρα να αρχίσουμε το επόμενο θέμα για την ε, ε, ομάδα δράσης για τον τουρισμό. Σας καλωσορίζω όλους. Δυστυχώς ο δεύτερος ομιλητής από το Λουξεμβούργο είναι στο τρένο. Και επειδή έγινε ένα δυστύχημα, καθυστέρησε το τρένο και δεν θα έρθει εγκαίρος. Οπότε θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη συνεδρίαση στο συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, θα ακούσουμε πρώτα το συντάκτη της ε, μελέτης ε, με θέμα βιώσιμος τουρισμός και ε, στατιστικές στο τομέα του τουρισμού. Την αναθέσαμε στη μελέτη και την παρακολούθησε το επιστημονικό μας τμήμα. Για διάφορους λόγους χρονικούς χρειάστηκε να αναβληθεί πολλές φορές η παρουσίαση και καλωσορίζω τον καθηγητή Πάουλ Πέτερς από το Πανεπιστήμιο της Μπρεντά στην Ολλανδία και μετά θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει πώς θέλει να εφαρμοστεί. Α, α όχι, αυτός είναι που λείπει. <laughs> Ζητώ συγγνώμη. Λέει κυρία Ταπαρδέλα, έχουμε πρόβλημα με τη διερμηνία από τα ρουμανικά. Βλέπω ότι οι συνάδελφοι διερμηνείς είναι εκεί και μιλούν, αλλά εμείς δεν τους ακούμε. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα υπάρχει με τα ρουμανικά. Ε, Τώρα είναι εντάξει. Λοιπόν, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Ισβανουή, αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας και αρμόδιο για την ομάδα εργασίας αυτή, για να μας ενημερώσει για τις πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες σε σχέση με τον τουρισμό. Το λόγο έχει λοιπόν ο Ισβαν Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι ως μέλος της Task Force ε, και ως πρόεδρος μάλιστα της ομάδας εργασίας ασχολήθηκα με τον τουρισμό στην Ευρώπη. Γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω μερικά λεπτά και αν θέλετε να με συμπληρώσετε, να με διορθώσετε, παρακαλώ να το κάνετε. Πριν από δύο εβδομάδες, στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, ψηφίσαμε για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχουμε επιτύχει μια μεγάλη στρατηγική νίκη σε συνεργασία και με το Λαϊκό Κόμμα. Κάναμε μια πρόταση, δηλαδή να ορίζεται κάθε χρόνο Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Τουρισμού. Έτσι, Ευρωπαϊκή Τουριστική Πρωτεύουσα. Αυτό ήταν μια δική μας πρωτοβουλία και βεβαίως χρειαζόταν να συμφωνήσει ε, και η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, η οποία και συμφώνησε. 2,5 ε, εκατομμύρια έχουμε εξασφαλίσει για να προετοιμάσουμε το σχέδιο αυτό την επόμενη τριετία. Εγώ ενημέρωσα όλους τους συναδέλφους και αν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα αυτό, παρακαλώ, βρίσκεται ε, και ο κύριος Κοράτσα. Ε, και το ιδιαίτερο γραφείο της ε, Επιτρόπου της ίδιας τα γνωρίζει αυτά τα θέματα και θέλει να τα προωθήσει. Χρειάζεται δηλαδή συνεργασία των διαφόρων θεσμικών οργάνων για να αρχίσει αυτή η προσπάθεια. Θέλω επίση να σας ενημερώσω ότι τις προάλλες ε, στο Λονδίνο συνεδρίασε μια ε, ομάδα ε, ευρωσυνικής συνεργασίας για τον τουρισμό. Ήταν μερικέ εκατοντάδε οι συμμετέχοντες σε αυτή τη διάσκεψη, παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Είναι μια δράση Ευρώπη-Κίνα, πάλι μετά από δική μας πρωτοβουλία της Επιτροπής μας, που έχει ξεκινήσει πριν από δύο χρόνια. Και μάλιστα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματα αυτά. Και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ε, αν θέλετε μπορείτε να έρθετε κοντά μας, μπορείτε να βοηθήσετε στην προσπάθεια αυτή. Όλα αυτά σας τα λέω εισαγωγικά και ενημερωτικά. Ο Γενικός Γραμματέας του Παγκοσμίου ε, Οργανισμού Τουρισμού θα έρθει στις Βρυξέλλες για διαπραγματεύσεις 6 με 8 Δεκεμβρίου. Συμμετέχω και εγώ σε αυτό το πρόγραμμα και σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε ή θέλετε να πείτε κάτι σχετικά, παρακαλώ μην διστάσετε. Έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε και να τα συμπεριλάβουμε. Τι άλλο να πω. Και πάλι με τη βοήθεια της Γραμματείας της Επιτροπής και της Ούρσουλα. Συμμετείχαμε στο φόρουμ για τον τουρισμό που έλεγε χώρα στην Πρατισλάβα και συζητήσαμε εκεί θέματα και της κοινοβουλευτικής μας ε, δραστηριότητας. Θα σας ενημερώσω γραπτός γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο αυτή τη στιγμή. Κάτι άλλο ακόμα ενημερωτικά για την ε, Επιτροπή Περιφερειών που είναι εδώ στο διπλανό κτίριο, είναι γείτονα. Ε, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με την Επιτροπή των Περιφερειών η οποία έχει καταρτήσει έκθεση για μέτρα περιφερειακής ανάπτυξης και εξετάζει και τις δήματα που μας ενδιαφέρουν. Και σε περίπτωση που χρειάζεστε πληροφορίες για τη δουλειά σας ή αν θέλετε να κάνετε κάποιες επαφές ε, με την Επιτροπή των Περιφερειών, έχουμε τη δυνατότητα και έχουμε και τα ονόματα ε, των ε, ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Και προγραμματίζουμε και άλλες κοινέ δραστηριότητες και συνεδριάσεις. Ο πρόεδρος Κράμερ ε, το τελευταίο διάστημα δραστηριοποιήθηκε πάρα πολύ και είχαμε και πολλές συζητήσεις για το πρόγραμμα Interrail. Θα το θυμάστε. Ε, για τους νέους, τους οποίους τα κάναμε δώρο για τα 18 γενέθλιά τους, ένα ε, πάσο Interrail δωρεάν. Εγώ διοργάνωσα ένα πρόγευμα εργασίας και κάλεσα δύο Γερμανούς ε, που είναι εμβληματικέ προσωπικότητες στην Γερμανία, δύο νέοι που το έχουν αναλάβει να το προωθήσουν αυτό. Και θα έρθει και ο πρόεδρος, αν ενδιαφέρεστε κι εσείς, επίκειται αυτό, δεν έχει γίνει ακόμα, ε, αξίζει τον κόπο, αν σας ενδιαφέρει είστε ευπρόσδεκτοι. Βέβαια, αυτό είναι θέμα μεταφορών, αλλά είναι θέμα και τουρισμού. Δύο πράγματα ακόμα. 15 Νοεμβρίου, το ξέρετε όλοι, το έχετε λάβει τις προσκλήσεις, γιατί ε, τις έστειλα την περασμένη εβδομάδα. Επίσης υπάρχει μια οργάνωση ε, από τον Ειρηνικό και την Ασία. Έχω ε, προσκαλέσει το Διευθυντή. Είναι μια εκδήλωση στο Λονδίνο προχτές. Εμείς ποτέ δεν είχαμε στο παρελθόν επίσημη ε, συνεργασία και επαφές ε, με αυτό το μεγάλο τουριστικό οργανισμό και θα πρέπει να καλύψουμε αυτό το κενό. Έρχονται λοιπόν υπουργοί από τις ασιατικές χώρες της Βρυξέλλες με τους οποίους πρέπει να έχουμε επαφές. Με τη γραμματεία επίσης θέλουμε να φροντίσουμε να έχουμε θέματα για τη συνεδρίαση της ειδική ομάδας της Task Force μέχρι το Δεκέμβριο για να προετοιμάσει κάτι για την επόμενη χρονιά ε, η γραμματεία. Και ένα τελευταίο σχόλιο, πάρα πολύ μικρό. Το 2017 καλό θα ήταν... Ε, ε, να μπορέσουμε να εορτάσουμε το έτος του βιώσιμου τουρισμού. Γιατί σε αυτό τον αστερισμό εγγράφεται το 2017. Και αν σας ενδιαφέρει παρακαλώ να το δηλώσετε συνεννοήθηκα με τον Γενικό Γραμματέα του της Παγκόσμιας Ένωσης Τουρισμού να στείλουμε κάποιους δικούς μας συναδέλφους, μέλη της Επιτροπής μας, στις συνεδριάσεις της δικές τους. Αυτά τα ολίγα και πάρα πολύ σύντομα. Είμαι στη διάθεσή σας. Έχουν έρθει και δήμαρχοι ε, από τις Κανάριες ε, νήσους. Τους έχει καλέσει η κυρία Γιάλα Σέντερ. Καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζουμε να περάσετε καλά. Είναι πολύ σημαντικός τουριστικός προορισμός τα Κανάρια νησιά στην Ευρώπη και είμαι βέβαιος ότι οι δήμαρχοι ε, θα αισθανθούν πάρα πολύ άνετα εδώ στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Ε, χαίρομαι που σας βλέπω. Το λόγο έχει ο καθηγητής Παουλ Πέτερς. Παρακαλώ. Okay, thank you very much, uh, Mr. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω αυτή τη μελέτη εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Βεβαίως δεν έχω συντάξει μόνος μου την ε, μελέτη από πολλές διαφορετικές πηγές, 7 τουλάχιστον, ε, συνεργαστήκαμε για να υποστηριχθεί η κεντρική μας ομάδα στο Μπρεντά. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να δούμε ποιες είναι οι τρέχουσες δραστηριότητες ε, στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού ιδίως τα προϊόντα που παρέχονται από το βιώσιμο τουρισμό σε αντιδιαστολή με τον ίδιο το βιώσιμο τουρισμό είναι διαφορετικά πράγματα. Μία εικόνα για να καταλάβετε Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος αλλάζει διαρκώς και διωγγώνεται Για το κλίμα λόγω χάρη, όσα προκαλεί η αεροπλοεία δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί. Επίση, τα προϊόντα βιώσιμου τουρισμού μπορεί να είναι ένα δρόμο για, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και φαίνεται να μην υπάρχει καλή αντιστοίχηση τουρισμού καθώ και περιβαλλοντικών αλλά και συγκοινωνιακών πολιτικών. Επίση, χρειάζεται παρακολούθηση που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει για τον βιώσιμο τουρισμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. So let's first look Ας δούμε πρώτα απ' όλα τις περιβαλλοντικές πτυχές. Θα τα βρείτε στη σελίδα 25 της μελέτης, τα έχετε και μπροστά σας. Υπάρχουν αρκετά περιβαλλοντικά ζητήματα σε σχέση με τον τουρισμό και τις ε, σχετικές μεταφορές. Το 2004 συντάξαμε μια έκθεση σχετική η οποία δείχνει ότι καθυστερούμε στο να παρακολουθήσουμε τα όσα συμβαίνουν. Αυτό που δείχνουν αυτοί οι αριθμοί είναι το εξωτερικό κόστος όλων αυτών των περιφερειακών θεμάτων, όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές, η ατμοσφαιρική ρήπανση, ο θόρυβος και το καθεξής. Αυτά επηρεάζουν τον ενδοευρωπαϊκό τουρισμό κατά 125 εκατομμύρια ευρώ ετησίω. Δεν είναι αμεληταίο το ποσό. Εάν ε, βάλουμε και τον εξωτερικό τουρισμό, τριπλασιάζεται το κόστο. Το βασικό κόστο το πληρώνουμε λόγω των κλιματικών αλλαγών. Ακόμα και αν είναι πολύ χαμηλέ εκτιμήσει, για το ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, είναι μεγάλο το περιβαλλοντικό κόστος. Πριν δούμε τα κοινωνικο-οικονομικά θέματα, κατά πρώτον, οι αριθμοί που δείχνω εδώ δείχνουν ότι ο τομέας του τουρισμού είναι ένας σημαντικός οικονομικός κλάδος. Είναι ένας κλάδος όπου το μεγαλύτερο μέρος των ταξιδιών γίνονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Και τα μισά τουλάχιστον είναι εσωτερικά ταξίδια και όχι διεθνή. Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο είναι η εποχικότητα των ε, εργασιακών θέσεων. Αυτό ασκεί πιέσεις στους εργαζομένους και καθιστά δύσκολο το να είναι καλές οι συνθήκες εργασίας. Βασίσαμε τη μελέτη μας σε συγκεκριμένα παραδείγματα με 162 συγκεκριμένα case studies που απαριθμώνται στο παράδειγμα της έκθεσης. οι οποίες προέρχονται από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, και αυτό που, καταλή... που ανα... είναι ότι οι περισσότερες περιπτώσεις, περισσότερες προσπάθειες βασίζονται στην κρατική χρηματοδότηση. Χωρίς αυτήν δεν μπορούν να συνεχίσουν. Και κάτι άλλο που έγινε προφανές είναι ότι δεν υπάρχουν ποσοτικές αξιολογήσεις για το περιβαλλοντικό και τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο. Δεν ξέρουμε τι συνέβη. Κάτι άλλο που ήταν σαφές είναι ότι οι περισσότερες περιπτώσεις που μελετήσαμε είχαν να κάνουν με το επίπεδο του προορισμού. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταφορές προ και από, στον, ε, από τον προορισμό δεν συμπεριλαμβάνονται. Περίπου 5 με 10 από τις περιπτώσεις μας συμπεριλαμβάνουν κάτι για τις μεταφορές. Ένα παράδειγμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταφορών. Τα μαργαριτάρια των Άλπαιων 25 προορισμοί στις Άλπεις που συνεργάζονται εδώ και πολλά χρόνια. Έχουν συνδυάσει τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν τους τουρίστες να έρχονται σε, ε, στους προορισμούς αυτούς με περισσότερο περιβαλλοντικά φιλικούς τρόπους. Και περισσότερη διασύνδεση μεταξύ των προορισμών αυτών ονομάζεται ήπια κινητικότητα. Είναι αυτή η νέα αρχή. Σε κάποια από τα μέρη αυτά είναι πετυχημένη όλη η προσπάθεια. Ακόμη και όσοι δεν έχουν σιδηροδρομικό σταθμό καταφέρνουν να προσελκύσουν τους επισκέπτες τους φροντίζοντας τα τελευταία χιλιόμετρα από τον ε, συγκεκριμένο τοπικό σταθμό να τον ε, διασυνδέσουν με λεωφορείο. 25 λοιπόν προορισμοί εδώ και χρόνια δεν μεγαλώνει η ομάδα αυτή, παραμένει μικρή. Γιατί είναι περίπου πάνω από χίλιοι προορισμοί στις ε, Άλπεις. Βεβαίω κοιτάξαμε και τις πολιτικές. Από την σκοπιά του τουρισμού και των βιώσιμων μεταφορών είδαμε ότι ο βιώσιμος τουρισμός και οι μεταφορές δεν είναι πάντοτε ευθυγραμμισμένοι μαζί με τις περιβαλλοντικές πολιτικές, οι οποίες κοιτάζουν περισσότερο ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέσο όρο της, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν κάποια από τα προβλήματα, όπως τις κλιματικές αλλαγές. Ενώ ο τουρισμός είναι πιο bottom-up Δηλαδή από κάτω προς τα πάνω προσπαθούμε να δούμε τι προβλήματα μπορεί να προκαλεί ο τουρισμός ε, στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Αυτό είναι δύσκολο όπως έχουν τώρα τα πράγματα και όπως σχεδιάζονται οι τουριστικές πολιτικές. Αυτή η γραφική παράσταση δεν υπάρχει στην έκταση αλλά βλέπετε μια αναφορά σε αυτό το πρόβλημα. Και βλέπετε την εξέλιξη του συνόλου των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στον κόσμο. Αυτές οι δύο διατεκομένες γραμμές που πηγαίνουν προς τα κάτω είναι αυτά που συμφωνήσαμε στο Παρίσι. Με την υπόθεση ότι η συμφωνία κυρώνεται και ακολουθούμε την πράσινη γραμμή. Η κόκκινη η, αναφορά, η γραμμή αυτή αναφορά όπως ονομάζεται είναι οι διεθνείς οι εκπομπές της αεροπλοίας μαζί με τα πρότυπα της, του ΙΚΑ όπως συμφωνήθηκαν το Σεπτέμβριο στο Μόντρελ και όπως βλέπετε στο δεύτερο μισό του αιώνα δεν θα καταφέρουμε τίποτα εάν δεν καταβάλουμε προσπάθειες από όλους τους τομείς μαζί. Αλλά αν ένας τομέας ρηπαίνει περισσότερο από ό,τι όλοι μαζί και δεν κάνει τίποτα, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Έτσι λοιπόν ο ΙΚΑΟ προβλέψει μέτρα ε, τα οποία είναι επικεντρωμένα στην αγορά. Δηλαδή η αεροπλοεία δεν θέλουμε να καλύψει το κόστος όλων των άλλων κλάδων. Γιατί για την ώρα αυτό κάνουν. Δεν μειώνουν τι δικέ του εκπομπέ, πληρώνουν και αυτές άλλων. Η κόκκινη λοιπόν διατεκομένη γραμμή σας δείχνει τι πρέπει να κάνουν οι υπόλοιποι. Ελπίζοντας ότι θα φτάσουμε σε αρνητικά επίπεδα το 2080. Η αεροπλοεία λοιπόν είναι ένα πρόβλημα αρκετά περίπλοκο που σίγουρα θα μας αποσχολήσει και στο μέλλον. Βεβαίω, μια ερώτηση είναι τι μπορεί να κάνει ο κλάδο του τουρισμού για αυτά τα θέματα. Μια από τι περιπτώσει που μελετήσαμε στην έκθεση είναι μια πρόσφατη Ολλανδική περίπτωση. Μια εταιρεία που ονομάζεται Καρμακόπ και ετοίμασε, έφτιαξε έναν υπολογιστή για, τον, για τις εκπομπές του άνθρακα που ονομάζεται Καρμακάλ με 25 περιπτώσεις μεταφορών για τις αερομεταφορές ε, εντοπίζεται κάθε ξεχωριστό συνδυασμός αερομεταφορέα με αεροσκάφος και βλέπουμε το αποτύπωμα άνθρακα της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Βεβαίως είναι ένα εργαλείο business to business από εταιρεία προς εταιρεία, οπότε οι χρήστες διευκολύνονται τρομερά και μπορούν να το δουν και όλες οι οργανώσεις του προορισμού. 500.000 όνομα, υπολογίζεται ότι είναι το αποτύπωμα άνθρακα όλων των εταιριών αεροπλές στην Ευρώπη. Πολλές από αυτές εδράζονται στην Ευρώπη. Και συμπεριλαμβάνονται και κάποιες από τις δραστηριότητες του τουρισμού που είναι πολύ εντατικές στην κατανάλωση άνθρακα. Αυτό μας ενδιαφέρει για, την, ε, ε, για το σχεδιασμό προϊόντων, αλλά και την παροχή υπηρεσιών στο επίπεδο των προορισμών. Αυτό με φέρνει σε κάποια βασικά συμπεράσματα. Έλλειψη ενημερωμένων ε, δεδομένων για τις κοινωνικές και επιπτώσεις του τουρισμού, μια ανάγκη θεώρησης προς το μέλλον, όχι μόνο ότι θα γίνει μέσα στον ορίζοντα μιας δεκαετίας, αλλά και παραπέρα. Υποδομές για σιδηροδρόμους, αεροπλοεία, αυτά που τώρα φτιάχνουμε, υπάρχουν, αλλά χρειάζεται και μια πιο διορατική στάση. Ε, επίσης, Οι πιο βιώσιμες πρωτοβουλίε που διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν βασίζονται στην ε, δημόσια κρατική επιδότηση και χρηματοδότηση. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη βιώσιμων πρακτικών. Οι πολιτικές για τον τουρισμό, το περιβάλλον και τις μεταφορές δεν είναι πάντοτε ευθυγραμμισμένες και οι αερομεταφορές παραμένουν ένα πρόβλημα περίπλοκο. δεν έχει επιληθεί παρά τις πρωτοβουλίες του ΙΚΑΟ. Κάποιες συστάσεις που εκπορεύονται από τα συμπεράσματά μας. Παραπέμπουμε και πάλι στα πολύ σωστά συμπεράσματα της μελέτης του 2004 για να δούμε το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο του τουρισμού στην Ευρώπη ξανά με ένα νέο βλέμμα. Ίσως επίσης χρειάζεται μια επαναστάθμιση ε, του καταλόγου των ε, προορισμών, των σημείων προορισμού και των προϊόντων του βιώσιμου τουρισμού ε, για να υπάρχει μια καλύτερα στοχευμένη πολιτική τουρισμού στην Ευρώπη και μετά πρέπει να δούμε τον αντίκτυπο των μεγάλων έργων μεταφορών σε σχέση με το βιώσιμο τουρισμό. Επίσης, για τις μεταφορές, τις τουριστικές μεταφορές, βασική ε, περιβαλλοντική μέρημνα αυτών θα πρέπει να είναι η κάλυψη της αεροπλοείας. Λόγου χάρη, το συνδεδομικό δίκτυο δίνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Εν μέρη, διότι οι αποστάσεις που διανύει βεβαίως καρύς με τρένο είναι πολύ μικρότερες κατά μέσο και πολύ συντομότερες. Είναι μεγάλη διάρκεια των πτήσεων που δημιουργεί πρόβλημα. Πρέπει να προσέξουμε να μην εξαρτηθεί περισσότερο από ότι τώρα ο τουρισμός από την αεροπλοεία. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και με τις τωρινές τάσεις θα συνεχιστεί η τάση να χρησιμοποιούν, θα, συνεχιστεί η συνήθεια να χρησιμοποιούν περισσότερο το αυτοκίνητό τους. Κανείς δεν καταλαβαίνει όμως πόσο ανατρέχουμε και στα αεροπορικά ταξίδια. Επίσης θα χρειαστεί δικαιότερος ανταγωνισμός μεταξύ των ε, μεταφορέων low cost καθώς και των σιδηροδρόμων λεωφορείων ε, πούλμαν. Για τους προορισμούς υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης του άνθρακα και οι αερομεταφορές θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα σχετικά συστήματα για να δώσουν τα απαραίτητα αποτελέσματα. Και για τις επιχειρήσεις ισχύουν περίπου τα ίδια. Υπάρχουν ήδη κάποια προγράμματα με οικολογικά σήματα. Είναι τόσα πολλά βέβαια που το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Να κάτι που θα μπορούσε να βελτιωθεί. Ως προς την κατάρτιση ακόμη υπάρχει δουλειά να γίνει. Και χρειάζεται και η πρόληψη εργαλείων για τους διαχειριστές του τουρισμού. Επίσης, κάποιες διαπιστώσεις για τη συζήτησή σας, αλλά νομίζω ότι ήδη έχω πει αρκετά, οπότε καλύτερα να κλείσω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας και τώρα μπορούμε να πούμε στη συζήτηση. Κλάδια Μοντέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να χαιρετήσω τον ε, καθηγητή και να τον ευχαριστήσω για αυτή την παρουσίαση, την παρουσίαση της μελέτης. Θα, δεν θα παραλείψω να συμφωνήσω με τον ορισμό που εδώ περιλαμβάνεται ως προς τον βιώσιμο τουρισμό που δεν είναι απλώς μία νύχη της αγοράς, ένα μερίδιο της αγοράς, αλλά μία κεντρική γραμμή που μπορεί να ακολουθήσει ολοκλήρως ο τουριστικός κλάδος και θα πρέπει να λάβει σάρκα και οστά, με συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές αποφάσεις που θα ληφθούν ε, σε πέδο κάθε προορισμού, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες ολόκληρου του κλάδου. Ως μορφή συμπληρωματικός τρόπος να στηρίξουμε τον βιώσιμο τουρισμό, Δεν πρέπει να ξεχάσουμε την έννοια του εφιούς τουριστικού προορισμού, του καινοτόμου τουριστικού προορισμού, που με τεχνολογικά μέτρα, με την ψηφιοποίηση θα ενισχυθεί και θα γίνει καθεστώς, για να έχουμε τη βιώσιμη διαχείριση προορισμών που θα καλύπτουν και τις ανάγκες των συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών, ως προς την προσβασιμότητα και την δυνατότητα κάποιοι προορισμοί να είναι προσβάσιμοι σε όλους, με ε, κάλυψη τοπικών αναγκών, αλλά και το εξή θέμα, με τις συστάσεις, βλέπουμε, στις συστάσεις μάλλον βλέπουμε να λείπει η σημασία της ψηφιοποίησης. Είναι μια μορφή για να βελτιωθούν όσα μας ανέφερε ο καθηγητής. Δηλαδή, ο κατακαιρματισμός μεταξύ τουρισμού, μεταφορών και περιβάλλοντος. Επίσης, μία ακόμη παρατήρηση. Έλλειψη δεδομένων για να καταλάβουμε και το ποσοτικό αντίκτυπο του τουρισμού στο περιβάλλον. Αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο, το θεωρώ πολύ σημαντικό να υπάρχει και αυτή η αναφορά για τις εργασιακές συνθήκες και έχοντας υπόψη ότι ο τομέας αυτός, ο κλάδος αυτός απασχολεί πάρα πολλούς νέους αλλά και γυναίκες και υπάρχουν πολλοί φραγμίους προς τις πολιτικές που σχεδιάζονται. Αυτέ τι δύο παρατηρήσει ήθελα να κάνω και να θέσω και δύο ερωτήσει. Η πρώτη για το ευρωπαϊκό σύστημα των ε, τουριστικών ε, εκπαιδευτών του έτης. Υπάρχει κάποιο feedback, υπάρχουν κάποιε αντιδράσει σε σχέση με του προορισμού ανακράτω. Όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρουμε να στηρίζει ακόμα αυτή την πρωτοβουλία. Εδώ πρέπει να δούμε αν ελήφθη αυτό υπόψη τη στιγμή σύνταξη τη μελέτη και τι αποτελέσματα υπήρξαν. Ε, και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να στηρίζουμε ακόμα αυτήν την ε, πρωτοβουλία για τις σχολές τουριστικών επαγγελμάτων. Ακόμη, αναφερθήκατε στις μεταφορές ε, στον τουρισμό και το 8% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Ε, νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μια σειρά από κίνητρα και στους υδροδρόμους και να μειώσουμε την εξάρτηση από την αεροπλοεία. Ε, σωστά είπατε ότι αυτά πρέπει να κάνουμε, όμως έρχομαι από περιοχή νησιωτική. Και η ερώτησή μου είναι οι νησιωτικές ε, περιοχές και τα κράτη με νησιά που έχουν με μόνη πρόσβαση ακριβώς ε, τους θαλάσσιους δρόμους, αλλά και τις αερομεταφορές. Τι να κάνουν για την πραγματικότητα αυτή πώς θα καλυφθούν στην πράξη ανάγκες αυτών των περιοχών. Ήθελα την άποψή σας σχετικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η Κλάουντα Ταπαρντέλ. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω πως είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που είχα την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα του βιώσιμου τουρισμού εδώ στη δική μας Επιτροπή, ε, δεδομένου ότι η επόμενη χρονιά, το 2017, είναι ε, και χρονιά του βιώσιμου τουρισμού σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ όπως και οι συνάδελφοι τον καθηγητή που μας παρουσίασε τη μελέτη αυτή. Όλο και οι περισσότερες περιφέρειες σήμερα προσπαθούν να αναπτύξουν τον τουρισμό τους. Και βέβαια αυτό έχει πάρα πολλές επιπτώσεις για το περιβάλλον και για τους ε, φυσικούς πόρους συμβάλλει δε στην μεγαλύτερη ρήπανση. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να προσφέρουμε τις λύσεις που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα και ίσως κάποιες λύσεις που θα ε, συνδυάζονται με την σφαιρική ε, στρατηγική της Ευρώπης για την καταπολέμηση της απειλής από την κλιματική αλλαγή. Όπως ξέρετε και εσείς συνάδελφοι, εγώ θέλω να στηρίξω το βιώσιμο τουρισμό στην Ευρώπη. Και μαζί με τους συναδέλφους έχουμε πετύχει πολλά. Θα ήθελα να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα στο γεγονός πως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώσαμε ε, μία εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού στην οποία συμμετείχαν και συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και δύο επίτροποι ε, των οποίων η εντολή καλύπτει θέματα σχετικά με τον τουρισμό. Δηλαδή ο κύριος Ναύρατσιτς και η κυρία Πιενκόφσκα. Εορτάσαμε λοιπόν ε, σε αυτή την εκδήλωση την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού αλλά ο βασικός στόχος ήταν να, να συναντηθούμε όλοι μαζί για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στον ευρωπαϊκό τουρισμό σήμερα. Να δούμε ε, τι γίνεται με τη βιωσιμότητα, ε, με τα υπόλοιπα θέματα τα οποία προκύπτουν και παράλληλα Πιστεύω πως ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να γίνει μεγάλη επένδυση στις υποδομές, στην πολιτιστική κληρονομιά, όπως επίσης και στο ανθρώπινο δυναμικό. Ας μην ξεχνάμε πως χρειάζεται επένδυση για να ε, διατηρήσουμε το φυσικό περιβάλλον και την κληρονομιά αυτή στην Ευρώπη. Και επειδή είχαμε τους ε, δύο επιτρόπους παρόντες στην ημερίδα μας, τόνισα την ανάγκη της ευρωπαϊκής στρατηγικής σχετικά με το θέμα αυτό, η οποία θα πρέπει να δώσει μια συνέχεια ε, στις τοπικές ε, πρωτοβουλίες, να τις συνδυάσει με κάποιες πρωτοβουλίες σε κεντρικό επίπεδο. Τώρα για τη μελέτη που παρουσιάσατε, μιλήσατε εσείς για βέλτιστες πρακτικές και για βιώσιμο τουρισμό. Στηρίζω πολύ θερμά τις συστάσεις που έχετε συμπεριλάβει στη μελέτη σας. Η ανάπτυξη ενός βιώσιμου τουρισμού σημαίνει πως θα πρέπει να βρούμε νέους τρόπους για να πείσουμε τον κόσμο να επιλέγει λιγότερο γνωστούς προορισμούς. Προορισμούς που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες. Και βέβαια επειδή είμαι Ρουμάνα θα μιλήσω για το Δέλτα του Δούναβη, γιατί ξέρετε πως πρόκειται για ένα μοναδικό οικοσύστημα με καταπληκτική ε, ποικιλία χλωρίδας και πανίδας και έχουμε τέτοιου είδους ε, φυσικά τοπία με τεράστιο δυναμικό. Θα πρέπει όμως να τα προστατεύσουμε, να τα προστατεύσουμε από τις επιπτώσεις του τουρισμού και θα πρέπει να στηρίξουμε και να προωθήσουμε προορισμούς στα πλαίσια του βιώσιμου τουρισμού, αλλά να δώσουμε και πρόσβαση στις περιοχές αυτές. Έτσι μπορούμε να κατευθύνουμε κύματα τουρισμού προς τις περιφέρειες αυτές. Όμως ας είμαστε προσεκτικοί. Και θα δώσω το παράδειγμα πάλι του δέλτη του, δέλτου του Δούναβη. Όταν μιλάμε για πλωτές μεταφορές θα πρέπει να είμαστε σίγουροι πως δεν επηρεάζεται πολύ αρνητικά το περιβάλλον, η χλωρίδα, η πανίδα ε, και στα ποτάμια και στις λίμνες που αποτελούν το δέλτα του Δούναβη. Ακόμα ένα σχόλιο. Και εδώ πρόκειται για μια περισσότερο γενική παρατήρηση που δεν συνδέεται τόσο άμεσα με τη συζήτηση της έκθεσης που κάνουμε σήμερα εδώ. Τα όσα είπε ο Ίστβαν προηγουμένως για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Τουρισμού. Ο κύριος Κοράντζα είναι εδώ σήμερα και νομίζω ότι εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρη για όλε τι λεπτομέρειε που συνδέονται με το project αυτό, αλλά θα ήθελα παρακαλώ στο μέλλον η τιμή αυτή του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Τουρισμού να μην αποδίδεται στις πιο γνωστές πόλεις που έτσι και αλλιώς υποδέχονται τεράστιες αριθμούς τουριστών αλλά να προωθήσουμε με την ευκαιρία αυτή πόλεις και κομμοπόλεις ακόμα που έχουν τεράστιο τουριστικό δυναμικό. Πόλεις που θα έπρεπε να γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες είτε για τα τοπία τους, είτε για το περιβάλλον τους, είτε λόγω πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουν. Και με τον τρόπο αυτό οι πόλεις αυτές, τα αστικά αυτά κέντρα θα γίνουν πιο γνωστά. και θα προσελκύσουν τουρίστες από όλη την Ευρώπη. Στο τέλος της θητείας μας θα ήθελα πραγματικά να υπάρχει ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού που θα συμπεριλάβει όλα αυτά τα θέματα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και τη βιωσιμότητα ευρύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Πίπερς για την ε, τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίασή του και την τόσο ωραία μελέτη που έχουν ε, πραγματοποιήσει στον Πρεντά. Είναι τόσα πολλά τα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε σήμερα εδώ. Όμως πραγματικά είμαι πολύ ικανοποιημένη που θα προωθηθούν λόγω χάρη γρήγορε υδροδρομικέ διασυνδέσει. Όπω εγώ που έρχομαι από την Ουαλία και μα ενδιαφέρει το δυναμικό που έχουμε για βιώσιμο τουρισμό να τα αξιοποιήσουμε. Έχουμε πρόβλημα μέχρι τώρα με τι διασυνδέσει μα. Καλό λοιπόν να υπάρξουν καλύτερε συνδρομικοί ε, κόμποι ε, και διασυνδέσει, ώστε να έχουμε μια ε, πιο μετα... ένα ευρυθμότερο σύστημα μεταφορών σε όλη τη χώρα. Και κάτι άλλο που, μιλήσα, που ήταν ε, οι τα πράσινα σήματα, οικολογικά σήματα, που είναι εκατοντάδες πλέον στην Ευρώπη. Κάποια είναι επιτυχή. Όμως μπερδεύουν τον κόσμο που μετακινείται από τη μια περιοχή στην άλλη μεταξύ χωρών. Διότι δεν υπάρχει ένα κοινό πρότυπο. Νομίζω ότι η ευρωπαϊκή επιστοποίηση για τις πράσινες αυτές, ε, για τα πράσινα σήματα είναι σημαντική. Το αναζητούμε και σε άλλου τομεί όπω το, τα τρόφιμα. Και εκεί έχει πετύχει. Να κάνουμε κάτι ανάλογο. Υπάρχουν επιτυχημένες τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες. Αναφέρατε το Παρίσι και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πιο ενημερωμένες μελέτες. Ξέρουμε περίπου που βρισκόμαστε, ξέρουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις του τουρισμού ε, στις κλιματικές αλλαγές, κυρίως με τις μεταφορές, όσες περισσότερες πληροφορίες βέβαια έχουμε τόσο καλύτερο, αλλά Θα πρέπει να δούμε θέματα όπως η διάβρωση, η υδάτινη πόρη και πραγματικά ποιε είναι οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών απευθείας στις τουριστικές επιχειρήσεις πώς μπορεί να δυσκολεύουν την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού. Και τελευταία μου παρατήρηση έχει να κάνει με τα κοινωνικά ζητήματα, τα κοινωνικονομικά, ζητήματα. Η βιώσιμη διαχείριση των ε, εργατικών δυνάμεων έχει να κάνει και με τον πολιτισμό και με τη γλώσσα. Εγώ εκπροσωπώ την Ουαλία. Ε, τα Ουαλικά σε κάποιες περιπτώσεις ε, είναι η βασική γλώσσα που χρησιμοποιείται στο τοπικό επίπεδο. Έχει λοιπόν σημασία αυτό και έχει σημασία και προ την κουλτούρα, τα πολιτιστική διάσταση, την πολιτιστική διάσταση του θέματος. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε λοιπόν την επίδραση του τουρισμού στις γλώσσες και τον πολιτισμό. Δεν είναι αρνητική αναγκαστικά, είναι εάν δεν αξιοποιηθούν σωστά οι επιδράσεις του τουρισμού, αλλά μπορούν να, ε, ε, αναλόγως οι διαφορές να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες των ανθρώπων από την επίσκεψη διαφορετικών τουριστικών προορισμών και περιοχών. Ευχαριστώ, Ενέσα Γιάννα Σέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον καθηγητή Πέτρας. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση της μελέτης. Να πω μερικά πράγματα. Πώς επιλέξατε τις χώρες αυτές. Ε, μελετήσατε περιπτώσεις, μελετήσατε με επισκέψεις και ποιες χώρες. Εμείς έχουμε πάει ακόμα παραπέρα, δηλαδή δεν είναι μόνο ο προορισμός, είναι το είδος του τουρισμού, θεματικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός ας πούμε, πολιτιστικός τουρισμός, έχει τεράστιες ε, συνέπειες. Ε, μπορεί να είναι να δεις μια πολιτιστική κληρονομιά ή να πας να δεις μια συναυλία ε, ένα συγκρότημα ροκ. Υπάρχει ο ιατρικός τουρισμός. Υπάρχουν λοιπόν θεματικές έτσι, ενότητες. Αλλάζει ο κλάδος και μετράμε τι αντίκτυπο έχουν συγκεκριμένα είδη τουρισμού και ποια θέλουμε να προωθήσουμε. Η Ισπανία φαίνεται ως δυτική χώρα. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε μεσογειακοί, αλλά εδώ μας έχετε κατατάξει στη Δύση. Γιατί μελετήσατε τον Ατλαντικό, βεβαίως ε, βρεχόμαστε και από τον Ατλαντικό και βρίσκονται και οι συνάδελφοι από τα Κανάρια ε, ως ζωντανή απόδειξη, αλλά είμαστε και μεσογειακή χώρα. Δεύτερον, Βλέπω ότι μελετήσατε κάποια ευρωπαϊκά έργα και έχετε επιλέξει το project EDEN, το οποίο έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΔΕΜ. Έχετε ξεχάσει όμως το πρόγραμμα Καλυψό, που είναι ε, κοινωνικό. Δηλαδή, να ξεφύγουμε από τη σεζόν, ε, τις υψηλές τουριστικές περιόδους Δηλαδή τα ξενοδοχεία ε, ξέρουμε ότι ερημώνουν και όλες οι δομές το χειμώνα ε, και ε, δηλαδή τα θέρετρα όλα αυτά είναι άδεια και μπορούμε να προωθήσουμε τον κοινωνικό τουρισμό για οικογένειες που έχουν δυσκολίες για να μην ρημάζουν οι τουριστικοί προορισμοί μας εκτός θερινής περίοδου. Πώς το έχετε σκεφτεί αυτό. Άλλο θέμα. Το θέμα Τώρα μιλάμε για την κυκλική οικονομία και εργαζόμαστε πολύ εντακτικά. Εδώ μιλάμε για, για υλικά και προϊόντα και αγαθά. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αγγίξουμε και τις υπηρεσίες. Δηλαδή, μια τουριστική υπηρεσία, μια προσφορά τουριστικής υπηρεσίας από το σχεδιασμό μέχρι την επιστροφή και τα συμπαραμαρτούντα στο σπίτι σου, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την κυκλική οικονομία. Δηλαδή, να μην έχουμε αρνητικές συνέπειες εξωτερικές. Πώς σας φαίνεται αυτό, θα μπορούσε να είναι σημαντικό στοιχείο για προβληματισμό. Μετά, αναφερθήκατε στις αερομεταφορές και συνάδελφος προηγουμένως. Ε, βεβαίως θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα νησιά και τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες ε, περιφέρειες. Δεν μπορούμε έτσι τυφλά να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει και ο τουρισμός με το σιδηρόδρομο, περισσότεροι με το αεροπλάνο μετακινούνται ε, οι τουρίστες και θα πρέπει να βρούμε και εκεί καινοτομία. Θέλω επίσης να μάθω ε, τι λέτε για τις στατιστικές ε, και τους αριθμούς. Μάλλον υπάρχουν κάποια τέλη που επιβάλλουν κάποιο φόρο ε, στον τουρισμό. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάζε τουριστών, ε, υπάρχουν χώρες που είναι οι χώρες προέλευση αυτών των τουριστών, όπου δεν είναι δωρεάν η πρόσβαση στην παραλία. Θες να πας στην πλάζ, κύριε, θα πληρώσεις για να μπει στην πλάζ. Ε, και τώρα που λέμε ότι μήπως βάλουμε τουριστικό φόρο και γίνεται χαμός με του tour operators. Δεν μπορούμε κάπως έτσι με έναν τρόπο πολιτισμένο να προωθήσουμε ένα τέλος τουριστικό και ε, έγινε μεγάλος λόγος για τον αντίκτυπο ε, ως προς τις ε, εκπομπές ρήπων. Υπάρχει κλιματική αλλαγή, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς επηρεάζει αυτή τον τουρισμό, γιατί υπάρχουν τουριστικοί προορισμοί που ήδη πλήττονται από την κλιματική αλλαγή. Ξέρω εγώ μπορεί να είναι περιφέρειες που εξαρτώνται από αυτή την ε, μόνο καλλιέργεια εντό εισαγωγικών έχουν μία οικονομική δραστηριότητα και αυτή είναι ο τουρισμό. Και με την κλιματική αλλαγή κινδυνεύουν ε, να τη χάσουν. Τι θα απογίνουν αυτοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα η Ισαμπέλα Δεμόντε. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Μπράβο και σε εσά και σε όσου εργάστηκαν ε, για την εικόνα τη εκθέση αυτή και στην Επιτροπή για την συνεισφορά του κυρίου Κοράτσα αφού επελέγει για να εργαστεί επί του θέματος. Βεβαίω αυτό που μας εκπλήσει στη μελέτη αυτή είναι ότι οι περισσότεροι τουρίστες που έρχονται από την Ευρώπη την ίδια αυτό μας παραπέμπει ακριβώς σε μια τάση που ήδη έχουμε μελετήσει και που μας οδήγησε στην εκπόνηση της έκθεσης της οποίας είμαι συγγετρία, δηλαδή το ότι δεν θα είμαστε πλέον ο πρώτος ε, παγκόσμιος ε, τουριστικός προορισμός. Ταυτόχρονα όμως είναι σημαντικό αυτό για να σκεφτούμε καλά τι πολιτικές θέλουμε να εφαρμόσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολιτικές ολοκληρωμένες, ενιαίες. Ο τουρισμός μας δείχνει ότι χρειάζεται ένα συσχετισμό με τις μεταφορές. Δεν μπορούν να είναι αδύναμες οι μεταφορές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Μόνο 4% ε, των τουριστών, α πούμε, καταφεύγουν στο τρένο. Δεν θα ήμουν τόσο απεσιόδοξη βεβαίω για τι αερομεταφορέ, διότι γίνονται πολλά. Γίνονται πολλά ω προ την χρήση εναλλακτικών ε, καυσίμων για την μείωση των εκπομπών άνθρακα και υπ' αυτήν την έννοια μπορούν να περιοριστούν οι εκπομπέ και οι ρήποι με καλύτερη επίση ε, διασύνδεση μεταξύ πτήσεων, άμεσων απευθεία πτήσεων και με τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Υπάρχει εδώ σχετισμό και με την υγεία. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην, ε, στον τουρισμό της υγείας, στον τουρισμό της ε, θεραπείας. Και αυτό θα πρέπει να ε, το αντιμετωπίσουμε, να το καλύψουμε, διότι είναι και αυτό ένα νέο μερίδιο της αγοράς, είναι μια νης της αγοράς, αλλά αυξάνεται διαρκώς για τον ε, βιώσιμο τουρισμό επίσης. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα εναλλακτικά καύσιμα στις μεταφορές. Κάτε με, οι υποδομέ υποδοχή κάνουν πολλά, όμω κάποιε φορέ γίνεται αυτό με τα δικά του μέσα και δεν καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν το κόστο. Θα πρέπει να το κόστος αυτό κάπως να περιοριστεί. Τι κάνουν λοιπόν ε, οι υποδομές υποδοχής για να μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, όπω ε, γνωρίζετε. Και για την ψηφιοποίηση, δεύτερη ερώτησή μου, η συνεργατική οικονομία μπορεί να είναι θετική θετικό στοιχείο αλλά και αρνητικό. Όσο οδεύουμε περισσότερο προς τη χρήση των σπιτιών από ότι των ξενοδοχείων υπάρχει από κάποια έννοια μια προστοχώρηση και ως προς τις μεταφορές, μεγαλύτερη χρήση των αυτοκινήτων ανταγωνισμό προ του σιδηροδρόμου, το τρένο. Εδώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω τι είδου προσέγγιση πρέπει να έχουμε, τι δεδομένα μπορούμε να συλλέξουμε ω προ την συνεργατική οικονομία για να υπάρχει ένα συνολικό πλαίσιο και να καταγράψουμε και τι τάσει που διαμορφώνονται με τα σχετικά δεδομένα. Ένα τομέα που αναπτύσσεται γοργότατα. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ε, προσεκτικοί για να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο και αυτού του ιδιαίτερου τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχετε ξανά την ευκαιρία να απαντήσετε σε όλα αυτά που ακούσατε κύριε Πέτρας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις και για όλα τα θέματα τα οποία θέσατε. Είναι αρκετά. Θα απαντήσω σε κάποια. Να σας πω καταρχήν πως ε, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δικτών για τον Τουρισμό γνωρίζουμε πως υπάρχει to get better I mean, it's... Και το χρειαζόμαστε για να έχουμε καλύτερα στοιχεία στη διάθεσή μας, για να δούμε δηλαδή ακριβώς ποιες είναι οι επιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη. Να δούμε δηλαδή τι συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα αυτό. Εθίχθηκε το θέμα του κατά πόσο θα χρησιμοποιούμε άλλα είδη συγκοινωνία και άλλα μέσα εκτός από τα αεροπλάνα και νομίζω ότι ενδεχομένως για αυτούς οι οποίοι είναι πιο απομακρυσμένοι ίσως, ίσως για αυτούς που είναι νησιωτικοί προορισμοί. Πρέπει να σας πω πάντως πως υπάρχει ένα θέμα το οποίο εκεί πρέπει να ληφθεί υπόψη, αλλά καταρχήν θα πρέπει να καταλάβουμε πως εάν αυτή τη στιγμή η, ο, κλάδος των αεροπορικών μεταφορών αναπτυχθεί με τον τρόπο που αναπτύσσεται και στηριχθεί από όλους τον κόσμο ε, όπως γίνεται σήμερα, ίσως μέχρι τα τέλη του αιώνα θα έχουμε 20 φορές, 20 φορές παραπάνω ε, αεροπορικό δυναμικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ενδεχομένως αυτό δεν χρειάζεται για να σωθούν κάποιοι νησιωτικοί προορισμοί. Ε, και αυτό ξέρουμε τι σημαίνει και για τη δράση που πρέπει να λάβουμε για την αλλαγή του κλίματος, μια και είναι ένα θέμα το οποίο πολλοί συζήτησαν. Δηλαδή, κλιματική αλλαγή, πώς επηρεάζεται από τον τουρισμό, ε, για τα χειμωνιάτικα αθλήματα για παράδειγμα. Ξέρετε τι συμβαίνει στις Άλπεις, που πολλές φορές είναι δύσκολο να έχεις λίγο χιόνι σε περιοχές που είχες παλιά πολύ. Για να είναι λοιπόν ισορροπημένη η εξίσωση αυτή, νομίζω είναι προ συμφέρον του κλάδου τέτοιου είδου θέματα κλίματο να αντιμετωπιστούν. Επίση, με ρωτήσατε τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Τουρισμού ότι δηλαδή αυτό δεν θα πρέπει να δίνεται ως τίτλος μόνο σε μεγάλες και πολύ γνωστές πόλεις και πρέπει να σας πω πως αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ευρωπαϊκό έργο που λέγεται Σκήτος που είναι η ε, υποδοχή που προσφέρει μια έξυπνη πόλη και πρέπει να σας πω ότι μια από τις πόλεις οι οποίες συμμετείχαν που είναι το Γέλτσεμπορκ στην Σουηδία που ακολουθούσαν μια στρατηγική marketing ε, για να γεμίσουν τα μικρά νησιά που έχουν κοντά στην ακτή τους και μετά από μια εκστρατεία ξεκίνησαν και την πρώτη μέρα αντιμετώπισαν τεράστιο πρόβλημα γιατί 10.000 άτομα κατέφτασαν στο νησί και όπως σας είπα είναι πολύ μικρό νησάκι και είχαν μόνο μία δημόσια τουαλέτα. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να δώσω λεπτομέρειες, παρά ήταν πετυχημένη η πρόθεση. Οπότε εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δηλαδή χρειάζεται μία ισορροπία μεταξύ δυναμικού και ανάπτυξης. Και αυτό να το θυμόμαστε. Λοιπόν, αεροπορικές μεταφορές, κλιματική αλλαγή, το είπατε πολύ συχνά και μία πρόταση ήταν να βρούμε εναλλακτικές, εναλλακτικά καύσιμα. Αυτό που γνωρίζουμε από τους επιστήμονες είναι ότι τα βιοκαύσιμα θα βοηθήσουν και είναι εύκολο να εφαρμοστεί γιατί απλώς θα αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα οπότε χρησιμοποιείς τους ίδιους κινητήρες, τα ίδια αεροσκάφη αλλά γενικά μειώνουν το αποτύπωμα του διοξιδίου του άνθρακα όχι στο 100% και κάποια ίσως αυξάνουν και το αποτύπωμα του διοξιδίου του άνθρακα οπότε ίσως εντείνουν το πρόβλημα οπότε αν είμαστε στο 30 με 60% καταλαβαίνετε πως το αποτύπωμα εξακολουθεί να είναι μεγάλο Βοηθάει λοιπόν, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Κάποιες μελέτες ασχολούνται με άλλου είδους εναλλακτικά καύσιμα, όπου όμως δυστυχώς χρειάζεται μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για να είναι πετυχημένα. Οπότε, κοιτάξτε, αν χρησιμοποιούμε ελληνική ενέργεια, είναι πολύ περιορισμένη στις